Ε, έλαβα γνώση της επιστολής που στείλατε στον πρόεδρο, εσείς ως πρόεδρος στην Επιτροπή του Προέδρου, ε, στην ε, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας. Συναντήθηκα με την, κυρία, με την της, επειδή είναι ασοσιέ η έκθεση, την κυρία Γκοντελίβε Γκβίστχουτ και καταλήξαμε σε μια συμφωνία όπως πράγματι ζητήσατε εσείς εκ μέρους της Επιτροπής. Αυτή η συμφωνία Διανημήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Άγρη και ίσως υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Δεν γνωρίζετε ότι έχει υποβληθεί ήδη χωριστές ψηφοφορίες, split votes, στα θέματα αυτά τα οποία αποτελούσαν και τις ενστάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και αναφέρομαι ότι θα υπάρχει χωριστές ψηφοφορίες στι παραγράφους 38, 39, 40, 43, 48, 53, 54 και 61. Θα υπάρχει χωριστή ψηφοφορία και split vote στην παράγραφο 47, στο πρώτο τμήμα, στο δεύτερο τμήμα και στο τρίτο τμήμα. Χωριστή ψηφοφορία στην παράγραφο 49, η οποία αναφέρεται στις σχέσεις, όπως είπατε πολύ σωστά, Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μερκοσούρ και, ε, στο, πρώτο τμήμα και στο δεύτερο τμήμα. Ε, ίσως ε, δεν λάβατε γνώση ότι αυτά έχουν ήδη κατατεθεί να υπάρχουν χωριστές ψηφοφορίε. Εγώ υπερασπίστηκα στην κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκω τη συμφωνία την οποία έκανα με την καλή συνάδελφο την κυρία Γκοντελίβετ Βίσχουτ. Άρα έχουμε δύο επίπεδα συνεννόησης. Το ένα είναι οι αρμοδιότητες και αυτές απαντήθηκαν με το αίτημα το οποίο εγώ υπέβαλα διαχωριστές ψηφοφορίες ανταποκρινόμενος σε αυτό που ζητεί η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου της οποίας μέλος είμαι και εγώ. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να προδικάσω πώς θα ψηφίσει ο ένας συνάδελφος ή ο άλλος στην Ολομέλεια. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο το λέω τώρα. Αυτά έχουν υποβληθεί ε, και έτσι θα ψηφίσουμε με χωριστές ψηφοφορίες σε ό,τι αφορά τα επίμαχα ζητήματα, σε ό,τι αφορά τι ενστάσει τι οποίε θέτει η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Και αυτό θέλω να γίνει απολύτω κατανοητό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. ναι, λέω ο γνωρίζω ότι υπάρχει αυτό το αίτημα για ψηφοφορία κατά τμήματα. Θα το συζητήσουμε στους συντονιστέ. Πάντως, θα ε, συνεχίσουμε το να έχουμε αυτό το δισκεδόν των αρμοδιοτήτων και δεν ξέρω κατά πόσον εμεί έχουμε τα θέματα της Άγκρη και η Άγκρη θα έχει τα δικά μας και θα, θα δεχθεί τις τροπολογίε. θα δεχτεί τροπολογίες ε, όπως δεχόμαστε εμείς επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε τη ζημιά γιατί έτσι είναι τα πράγματα τη αρμοδιότητα. Ε, είναι σωστό που θέτεται το θέμα αυτό και όχι μάλιστα μόνο στους συντονιστές αλλά και στα πλαίσια της δημοσίας ε, συνεδριάσεως. Και αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου είναι σωστά. Δεν μιλούμε για ένα πρόβλημα μονάχα σε τούτην την έκθεση, αλλά για ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται ξανά και ξανά. Η κυρία Μουσκαρδίνη είπε για άλλη επιτροπή, όπου ήταν η θέμα επισήμανσης ε, υφαντουργικών προϊόντων και αλλού σε άλλες εκθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα εμφανίζονται τροπολογίες επί ενός φακέλου που εμείς είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας. Εγώ πάλι τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο ημέρες ήμουν άρρωστο στο σπίτι, είχα χρόνο λοιπόν και μπόρεσα να εξετάσω προσεκτικά το σχέδιο εκθέσεως της κυρίας Κουίστχαουτ Ρόβολ. Εξέτασα λοιπόν τι ε, ψήφισε η Επιτροπή μας και ήταν ακριβώς σύμφωνα με τις διατάξεις. Κοίταξα και το σχέδιο εκθέσεως στην Επιτροπή Γεωργίας του κ. Παπαστάμκου και αυτό ήταν ακριβώς μέσα στα πλαίσια. Τώρα συνέβη το εξής. Στην Επιτροπή Γεωργίας κατατέθηκαν τροπολογίες οι οποίες είναι αντίθετες με τη συμφωνία. Και λέω εδώ καθαρά, κοιτάξτε, διαρωτώ εάν τέτοιες ε, εκβάσεις ψηφοφοριών είναι συμπτωματικές ή, ή αν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο. Γιατί υπάρχουν από καιρό τα έγγραφα αυτά και διαρωτώ με πώ, και το θέτω βέβαια κάπω επιθετικά, η γραμματεία τη Επιτροπή μα μετά την ψηφοφορία έρχεται και μα λέει υπάρχει ένα πρόβλημα, πράγματι συνέβη αυτό. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν πριν από την ψηφοφορία να εξετάσει η γραμματεία τη Επιτροπής τι έχει πει η Επιτροπή Γεωργίας για το άρθρο 50 και γιατί δεν βρίσκεται ένας τρόπος επιτροπές οι οποίες είναι εν κινούνται αντίθετα με τη συμφωνία για τις αρμοδιότητες των επιτροπών του άρθρου 50 να εμποδίζονται. Εγώ θέλω στο μέλλον σε μελλοντικά θέματα να είναι πιο προσεκτική η γραμματεία της Επιτροπής μας και δυνατόν να μας λέει πριν από τις ψηφοφορίες άλλων επιτροπών και να μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με άλλους συναδέλφους άλλων επιτροπών για να δούμε πώς να λυθεί το πρόβλημα. Πάντως εγώ κατ' επανάληψη έχω νευριάσει διότι δεν μας επέτρεψαν να ψηφίσουμε σε άλλες επιτροπές τροπολογίες διότι δεν ήταν παραδεκτές. Και διαρωτώ γιατί δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο, διότι τότε δεν θα είχαμε το πρόβλημα. Τώρα για το πρόβλημα την επόμενη εβδομάδα και μιλώ μόνο εξ ονόματος της ομάδας μου, θέλω να ψηφίσουμε την έκθεση του κ. Παπαστάμκου την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι εκ νέου παραπομπή στην Επιτροπή Γεωργία δεν θα προσφέρει απολύτω τίποτε. Θα προκαλέσει μονάχα αναβολή τη συζητήσεω αλλά του θέματο και τίποτε άλλο. Και η παράκλησή μου προ όλε τι ε, πολιτικές ομάδες είναι να εξετάσουμε ήρεμα, χαλαρά το σχέδιο που έχει υποβληθεί και να ξανασκεφτούμε εάν έχει όντως νόημα να μην είναι αρμόδια εξουσία η Επιτροπή μας αλλά η Γεωργική για θέματα που δεν είναι θέματα της αρμοδιότητάς μας και για το θέμα Μερκοσούρ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο θέμα των γεωργικών προϊόντων του Μερκοσούρ και θα ήθελα πολύ η Επιτροπή Γεωργίας να μας δώσει μια λίστα προβλημάτων από την ε, γεωργική σκορπιά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στις διαπραγματεύσεις. Θα ήταν λάθος να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ και αν δούμε μάλιστα και την αιτιολόγηση επειδή δόθηκε η εντολή πριν να συμπεριληφθούν ορισμένες χώρες ε, τότε θα πρέπει να διακόψουμε και τον γύρο Ντόχα που ασφαλώς έγινε, άρχισε δηλαδή πριν από την ε, διεύρυνση του 2004 και του 2007. Θα έπρεπε επίσης να διακόψουμε τι διαπραγματεύσει με την Κροατία γιατί άρχισαν πριν από το 2004 τις ε, ενταξιακές διαπραγματεύσει τη Τουρκία και ούτω καθεξής. Δηλαδή ένας ολόκληρος αριθμός διαπραγματεύσεων που έχουν αρχίσει πριν από 6-7 χρόνια. Και γι' αυτό εκνευρίζομαι με αυτή την περίεργη αιτιολόγηση γιατί δήθεν πρέπει να διακόψουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ. Ας το επανεξετάσουμε, ας έχουμε την δυνατότητα να ζητήσουμε ψηφοφορίε κατά τμήματα split votes και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα υποφερτό αποτέλεσμα. Για το μέλλον πάντως θα ήθελα πρώτα να μην αναπεμφθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή η έκθεση, αλλά ψηφιστεί. Και δεύτερο, η γραμματεία της Επιτροπής μας να ασχοληθεί πολύ εντατικότερα να ελέγχει πριν από τις ψηφοφορίες άλλων επιτροπών που ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος να ψηφιστούν τροπολογίες σε άλλες επιτροπές οι οποίε θίγουν τις δικές μας αρμοδιότητες και αυτό να αποφευθεί. Θα είναι καλό να προσπαθήσουμε εμείς ως Ευρωβουλευτές να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι, είναι πολιτικό το θέμα, αλλά είναι ταυτόχρονα και διαδικαστικό. Το τι να κάνουμε. κατόπιν της εγκρίσεως των τροπολογιών στην Επιτροπή Γεωργίας. Any Έχουμε τίποτα άλλο το ίδιο θέμα, κάτι διαδικαστικό. Θα, τα, θα το δούμε με τους συντονιστές. Το πολιτικό όμως θέμα θα πρέπει να το συζητήσουμε εδώ. Οπότε, έχετε κάτι άλλο, όχι. Εντάξει. Άρα το θέμα είναι σαφές. Πάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχετε έτοιμες τις κάρτες σας. Αρχίζουμε. Θα ψηφίσουμε τώρα ε, το θέμα, το, το, την έκθεση για τον κανονισμό όσον αφορά τις ε, γενικευμένες προτιμήσεις. Uh, Τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματο γενικημένων δασμολογικών προτιμήσεων ε, για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2009 31 Δεκάτου του 2011. Έχουμε εδώ μια σειρά από τροπολογίε ε, από την Επιτροπή Αναπτύξεως. Τώρα έχουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες εξελίξεις στο θέμα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, έχετε το λόγο κύριε Σόλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, θέλω να προβώ σε κάποια σύντομη δήλωση πριν αρχίσουμε τη ζωοφορία για την εκθεσή μου. Επανειλημμένα έχει συζητηθεί το ζήτημα το ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια ταχεία λύση όσον αφορά ε, αυτού του είδους την εφαρμογή του συστήματος των ειδικευμένων προτιμήσεων γιατί οι επιλέξιμες χώρες χρειάζονται ασφάλεια δικαίου, χρειάζονται ε, μια, μια κρυστάλλινη κατάσταση όσον αφορά την συνέχιση του συστήματος. Και επανειλημμένα έχουμε επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί νέα εκδοχή του νέου κανονισμού δεν την έχει εγκαίρως παρουσιάσει. Και αυτό προσπάθησα να εξηγήσω στο κείμενό μου. Ότι το Κοινοβούλιο Δυνάμει της τη Λισαβόνας έχει αρμοδιότητες συναπόφασης και εν προκειμένου. Είχαμε κάποιες εξελίξεις τελευταίες εβδομάδες, οπότε και ήρθα σε επαφή τους και οδείς και τους ευχαριστώ για την συνεργασία τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επιτέλους να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σε όλες τις φάσεις εξέλιξης ενός θέματος μιας ενός νομοθετήματος και έτσι το Κοινοβούλιο να μπορεί να λάβει υπόψη τις εξελίξεις. Καλώς όρισε και ο κύριος Επίτροπος στη σημερινή μας συνάντηση. Παρακαλώ να μας πει, αν θέλει, ότι και αυτός θα συμβάλλει στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε επίσης και την επιστολή του Γενικού Διευθυντού του Αρμοδιού, ο οποίος εξηγεί την πολιτική, τη στάση της ε, Επιτροπής της Περιπτώσεις. Έγινε ανταλλαγή των απόψεων στην ε, αρχή με το αρχικό κείμενο και είχαμε πει ότι ε, θα αναζητηθεί μια λύση όσον αφορά το δικαίωμα στην πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και ότι αυτό θα ενσωματωθεί στην περίπλοκη διαδικασία της συναπόφασης ε, και όσον αφορά τον μηχανισμό. Οπότε, κατόπιν αυτών των επαφών, εγώ απέσυρα όλε μου τι τροπολογίε, γιατί τηρώ τα συμπεφωνημένα ούτω και έτσι νομίζω ότι λύνεται το πολιτικό θέμα που έχουμε με την Κομισιόν. Και έτσι νομίζω ότι γέρος θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κάποια λύση για να εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός και αυτό θα ωφελήσει όλους και τις επιλέξιμες χώρες αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι κατανοώ πλήρως τις τροπολογίες της ΔΕΒΕ. Δυστυχώς οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα να αναζητηθεί μια λύση με την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Διότι η ΔΕΒΕ ήδη είχε προβεί στην ψήφιση και σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να ανακληθεί αυτή η γνωμοδότηση. Οπότε και εγώ έχω να σας πω ότι για τον ε, μηχανισμό των γενικημένων προτιμήσεων Είπαμε ότι θα έχουμε εξελίξει τον Μάιο, θα προσθεστεί τότε το νέο σύστημα. Και άρα θα προλάβουμε υπόψη τη γνώμη της ΔΕΒΕ. Και θα πούμε και τη δική μας γνώμη βέβαια, λαμβάνοντα υπόψη την νομική βάση που ήταν ε, η δική μου αφετηρία, ε, το πνεύμα που διαπνέει την εκθεσή μου. Γι' αυτό είπαμε να γίνει ψήφιση ε, όλων μαζί των τροπολογιών της ΔΕΒΕ. Εγώ τι θεωρώ θετικές αλλά λόγω της πολιτικής και τεχνικής, τεχνοκρατικής αποφάσεως που πρέπει να πάρουμε, σας ε, προτείνω να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, όπως προείπα. Πρόεδρος. Επομένως, θα κάνω αυτό που λέει ο εισηγητής. Και εγώ είμαι και ο εισηγητής και το έχουμε συζητήσει. Ο, οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και καθυστέρηση θα παραβλάψει τις επιλέξιμες χώρες. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε λοιπόν επειδή ήταν το λεγόμενο ρολόβερ δεν υπήρχε χώρος ε, να συζητηθούν ουσιώδεις τροποποιήσεις Επίσης κατανάθεση πράξεις μπορούν μείνουν στον κανονισμό Omnibus 1 και 2 που πρόκειται να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο από την Κομισιόν προσεχώς και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτά τα σχέδια πρωτοβουλειών θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας Επίσης, οι δικές μας τροπολογίες σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωση του Κοινοβουλίου από τούδε σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ως έχει, είναι εγγυημένες. Με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μου έχουν στείλει αναλαμβάνοντας δέσμευση, πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Και ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές θεώρησαν τις εν λόγω εγγυήσεις επαρκής για το θέμα αυτό, για τον φάκελο αυτό. Γι' αυτό και συμφώνησα με την απόσυρση των τροπολογιών μας και για τις τροπολογίες της ΔΕΒΕ Η δική μας πάντως αξιολόγηση της ουσίας των τροπολογιών αυτών που θα ληφθούν υπόψη όταν θα έρθει ο ουσιαστικός κανονισμός και θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για να εγκριθεί το σχέδιο κανονισμού ως έχει προταθεί από την Κομισιόν υπό τον μοναδικό όρο ότι θα μας εξασφαλίσουν ότι από τούδε η Κομισιόν θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο για κάθε βήμα σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Νομίζω ότι ήταν θετική η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ και τον κύριο Σόλτς και την Κομισιόν για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να οδηγηθούμε σε αίσιον πέρας. Ας προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες που προέρχονται από την Επιτροπή Αναπτύξεως. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία επί της τροποποιηθήσης προτάσεως Κομισιόν, ψήφι υπέρ. Άμεση χωρίτε πρόκειται για ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή με κάρτες, αρχίζει. Πέρας, ομόφωνα, ψήφος, ψηφοφορία τώρα επί του σχεδίου ε, νομοθετικού περιεχομένου, ψήφ... μάλλον πάλι, πάλι ονομαστική εδώ, λειτουργεί, λειτουργεί το μηχάνημά σας, κυρία Μουσκαλίνη. Ναι, έχουμε σημειώσει την ψήφο σας. Την έχουμε υπολογίσει. Πέρας τώρα της ψηφοφορίας 22 ψηφίσαντες 22 ψήφοι υπέρ. ομοφωνία λοιπόν. Συγχαρητήρια στον κύριο Σόλτς για την εξαίρετη εργασία. Και θα προχωρήσουμε τώρα στο υπαριθμόν 6 σχέδιο γνωμοδοτήσεως για την Επιτροπή ΙΜΚΟ επί της δικής τους το, ε, ε εκθέσεως για νέα αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Έχουν κατατεθεί 7 τροπολογίες. Θα προχωρήσουμε στις ε, τροπολογίες αυτές ξεκινώντας με την υπαριθμόν 1 ψήφι υπέρ κατά απογές εγκρίνονται εγκρίνεται μάλλον συμβιβαστική τροπολογία 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 με ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα της τροπολογίας 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 ψηφοφορία κατά τμήματα, τμήμα 1 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται Δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 30 λέει ο πρόεδρος τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται 33 κατά τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 συγγνώμη 34 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με συγχωρείτε ήταν κατά τμήματα πρέπει να επαναληφθεί 35-1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ας γίνει επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της 35 ε, ανοίγει η ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Λείπει κά, κάποιος. Ωραία, πέρασε. Απορρίφθηκε λόγω ισοψηφίας. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 κατά τμήματα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νέα τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κάποιος διακόπτη λέτε όλες μαζί δεν έχει κανένας ένσταση καλά λοιπόν μέχρι την 47 42-47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τελική ψηφοφορία ονομαστική ονομαστική αρχίζει Πέρας, το δε αποτέλεσμα είναι 17 υπέρ, ουδεμία ε, κατά και 5 αποχές. Συγχαρητήρια, Χωσέφα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι συνεργάστηκαν και τα πρόσωπα της Γραμματείας καθώς και άλλοι συνεργάτες το Λαϊκό Κόμμα, οι Φιλελεύθεροι, η Γκουε, η Πράσινη υπήρξε γενική συνεργασία, γενική συνένεση και είναι σημαντικό για να δοθούν ορισμένες σημαντικές κατευθύνσεις για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Μάλιστα, στο 7 τώρα εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά Έχετε κάποιο πρόβλημα με την μετάφραση, κύριε Μάρτιν. Μα τα λέω αγγλικά. Α, από τα ισπανικά μάλιστα. Λοιπόν, εμπορικές σχέσεις ενώσεως Καναδά. Πρόκειται για εξέταση ερώτησης με έτοιμα προφορικής απάντησης οι πολιτικές ομάδες είχαν συμφωνήσει επί μιας ταχείας διαδικασίας για την προφορική αυτή ερώτηση διότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε να δοθεί έγκαιρα έστω και ανεπίσημα απάντηση από την Κομισιόν για την σύνταξη του σχεδίου ψηφίσματος εν ώψη επίσκεψης της αντιπροσωπείας μας, της Επιτροπής μας δηλαδή στον Καναδά έχει συμφωνηθεί το σχέδιο από τις πολιτικές ομάδες από έξι πολιτικές ομάδες ώστε πρώτα πρέπει να δούμε εάν θα ψηφίσουμε αμέσως ή εάν θα δώσουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Δεν υπάρχει ένσταση να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία κύριε Κασπαρή. Όχι, ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στην ψηφοφορία του σχεδίου προφορικής ερωτήσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εμπορικές σχέσεις Ευρω... Ευρωπαϊκής Ενώσεως Καναδά όπως έχει περιβληθεί τον ε, τύπο συμβιβαστικού κειμένου από διάφορες πολιτικές ομάδες. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία που είναι ονομαστική. Πέρας. 19 ψήφοι υπέρ επί 19 ψηφισάντων. Ας προχωρήσουμε εδώ. Εδώ τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Προχωρούμε στο θέμα υπαριθμών 8. Υπάρχει μάλλον μια παρανόηση σχετικά με τον τίτλο, διότι πρόκειται στην πραγματικότητα για ενημέρωση από πλευρά του Επιτρόπου Ντεγκούχτ για θέματα σχετικά με την εμπορική διάσταση του κανονισμού νέων τροφίμων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία συνδιαλλαγής και η τελική συνεδρίαση θα γίνει 16 Μαρτίου με θέματα τροφίμων που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους. και τις σχετικές επιπτώσεις στο εμπόριο. Θεώρησα λοιπόν ότι δεν υπάρχουν υπάρχουν εμπόδια να μας ενημερώσει ο Επίτροπος για τις εμπορικές διαστάσεις του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Επειδή όμως ο κανονισμό βρίσκεται στην διαδικασία συνδιαλλαγής και μάλιστα στι τελικέ φάσεις, δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα να γίνει συζήτηση χωρίς παρέμβαση επί τη διαδικασία συνδιαλλαγή. Είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θα δώσω τον λόγο αμέσως στον Επίτροπο κύριο Ντεγκούχτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Προσήλθα σήμερα εδώ για να επιστήσω την προσοχή σας στην εμπορική διάσταση του σχεδίου κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες της Ευρωβουλής για θέματα κλωνοποίησης, κυρίως ηθικού χαρακτήρα, αλλά παραμένουμε στα πλαίσια του δικαίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τα όσα κάνουμε εδώ, με στην Ευρώπη, ωστόσο είναι δική μας υπόθεση. η απαγόρευση της κλωνοποίησης για παραγωγή τροφίμων μπορεί να ε, δικαιολογηθεί σύμφωνα με διατάξεις του ΠΟΕ, δεν έχει χαρακτήρα διακρίσεων και ούτως ή άλλως έχει και σημαντική επίπτωση στην υγεία των ζώων. Τουλάχιστον μέχρι ότου βελτιωθεί η τεχνολογία κλωνοποίησης. Από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι η απαγόρευση τροφίμων, ε, εισαγωγής τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα του απογόνους τους είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί. Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τις ε, συμφωνίες SPS που απαιτεί επιστημονική θεμελίωση επιστημονική θεμελίωση που έχει κάνει η ΕΦΣΑ δεν φαίνεται να εντοπίζει ανησυχίες που δικαιολογούν απαγόρευση εισαγωγών ούτε από την άποψη της ε, προστασίας των ζώων ε, για τους απογόνους, διότι ε, οι απόγονοι των κλωνοποιημένων ζώων εκτρέφονται με τις συνήθεις παραδοσιακές μεθόδους. Τα υπόλοιπα δεν υπάγονται στις συμφωνίες SPS Επίσης τονίζω ότι η εισαγωγή συστήματος προεγκρίσεως αγορών θα σήμαινε κάτι ταυτόσιμο με απαγόρευση. Εφόσον είναι ασφαλής η κατανάλωση προϊόντων απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, οποιαδήποτε καθυστέρηση η απαγόρευση εισαγωγής θα είναι αντίθετη με διατάξεις της Συμφωνίας SPS. Απαγόρευση η πρώτερη έγκριση εισαγωγών που καταλήγει σε de facto απαγόρευση της εισαγωγής από τρίτες χώρες επειδή οι χώρες αυτές δεν έχουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα τροφίμων για τρόφιμα που προέρχονται από απογόνους χρονοποιημένων ζώων θα σημάνει στην πράξη ότι θα σταματήσουμε τις εισαγωγές από τρίτες χώρες όπου γίνεται κλωνοποίηση η επιβολή απαγόρευσης αγωγής επιπροϊόντων απογόνων κλωνοποιημένων ζώων θα σημαίνει ότι ε, απαγορεύονται όλες αυτές τις αγωγές και οδηγούν σε μέτρα αντιπίνων. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, Πολιτείες, τα αντίπεινά τους θα μπορούσαν να είναι να καταγγείλουν την συμφωνία για τις ορμόνες και να αρχίσουν οι ε, κυρώσεις τύπου καρουσέλ και μπορούν να μας κοστίσουν αυτά 250 εκατομμύρια ε, ευρώ τον χρόνο. Το ίδιο μπορεί να τεθεί ως θέμα και για τους τροποποιημένους γενετικά οργανισμούς καθώς και για το κρέας πουλερικών. Λοιπόν, ε, το θέμα αυτό μπορεί να μας βάλει σε πολύ δύσκολη θέση. Όπως είναι προφανές, ο Επίτροπος αναφέρεται στην εμπορική διάσταση του θέματος και τον ευχαριστώ που ενημερώνει την Επιτροπή Εμπορίου με τις πληροφορίες αυτές. Έχοντας λάβει υπόψη τα όσα είπα πριν από την παρέμβασή του, θα δεχθώ ερωτήσεις μονάχα που θα έχουν ως στόχο διευκρίνηση των όσων δήλωσε ο Επίτροπος. Δεν θα επιτρέψω ερωτήσεις, μάλλον συζητήσεις επί της ουσίας. Φιέλνερ στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα εισέλθω στη συζήτηση. Είμαι μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας Τροφίμων κλπ. Έχω λοιπόν τη δυνατότητα να συζητήσω ε, το θέμα αυτό σε εκείνο το πλαίσιο. Αλλά για λόγους διαφάνειας θα ήθελα να ενημερώσω τα παρόντα μέλη ότι επί του παρόντος στην διαδικασία συνδιαλλαγής είναι σαφές ότι το Συμβούλιο μοιράζεται την γνώμη που εξέφρασε ο Επίτροπος για τα θέματα που συζητούμε τώρα και μου φαίνεται ότι εκεί είναι και το ζήτημα που περιπλέκεται η συζήτηση. Ευχαριστώ πάντως τον Επίτροπο που μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε διότι όταν βρισκόμαστε σε συζητήσεις στην συνδιαλλαγή είναι προφανές ότι εκεί εκπροσωπούνται ιδίω τα συμφέροντα της Επιτροπής η οποία συμμετέχει στην συνδιαλλαγή ενώ αυτό που έχει ειδικό σημαντικότερο ενδιαφέρον είναι να ε, προβληθούν τα συμφέροντα όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όπως είπε ο ίδιος ο Επίτροπος, με είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο θα υπάρξουν επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα δώσω τον λόγο μόνο σε μέλη της ε, Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Η κυρία Μουσκαρδίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο και για τη συνάντηση αυτή και για τα νέα τα οποία μας έδωσε. Θα ήθελα κάποιες ε, περισσότερες πληροφορίες για τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος. Αν ε, επί παραδείγματι γνωρίζουμε ότι απαιτούνται κάποια χρόνια προκειμένου να θεωρούνται έγκυρα τα πρωτόκολλα τα οποία φορούν ε, φαρμακευτικά προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που χορηγείται σε έναν οργανισμό. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι αυτά τα πρωτόκολλα μέσω των οποίων καθορίζεται ότι τα επιστημονικά στοιχεία είναι καθησυχαστικά για την ε, χρήση ε, τροφίμων που ε, προέρχονται από κλωνοποιημένα προϊόντα. Μας μίλησε ο Επίτροπος και για ένα δυνητικό πρόβλημα με τρίτες χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μέτρα κατά των δικών μας. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις για πιθανό κόστος ε, στην υγεία για ε, προϊόντα τα οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί και δεν έχουν εγκριθεί εδώ και χρόνια. Και τρίτον, κατά πόσο έχει αξιολογηθεί τι επιπτώσεις μπορούμε να έχουμε από οικονομικής πλευράς ε, εάν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα για τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα εάν δοθεί το πράσινο φως για την εισαγωγή ζώων ή οργάνων ζώων τα οποία εκτρέφονται ε, ή ακόμα και αν εκτρέφονται με παραδοσιακό τρόπο παράγονται κατά τρόπον ο οποίος αποκλίνει από τον παραδοσιακό. Εάν, για παράδειγμα, δίνονται γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί στι στις ζωοτροφές ε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μείωση στο κόστος ε, για την ανατροφή ζώων και τι κόστος μπορεί να υπάρχει για τις υποανάπτυκες χώρες. Μήπως παίρνουμε απλώς προϊόντα από χώρες οι οποίες δεν είναι κατάλληλα ανεπτυγμένες απλώς για να εξοικονομήσουμε χρήματα και όλα αυτά γίνονται εις βάρος της ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τέλει έχει λάβει υπόψη τις τι αρνητικές επιπτώσεις. Μπορείτε να μας δώσετε και κάποια επιπλέον ε, στοιχεία και επιστημονικά αλλά και συνολικά ως προς το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις τώρα προς τον Επίτροπο, David Martin. Δηλαδή συνεχίζονται οι ερωτήσεις προς τον κύριο Επίτροπο. Ευχαριστώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος δύο φορές και το Κοινοβούλιο δύο φορές έχει ξεκαθαρίσει με σημαντική πλειοψηφία ότι τα κλωνοποιημένα ζώα δεν πρέπει να εντάσσονται στην ε, αλυσίδα διατροφής. Θα υπάρξει ισοσύγκρουση με τον ΠΟΕ, αλλά και η προστασία ζώων και η αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη, εν πάση περιπτώσει, και άλλωστε η ασφάλεια δεν έχει ε, η ασφάλεια των σχετικών τροφίμων δεν είναι αποδεδειγμένη. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα σε τρίτες χώρες εταίρους δεν υπάρχει σύστημα εχνηλασιμότητας για τα προϊόντα το επιχείρημα λέει ότι θα πρέπει τότε να απαγορευτούν όλε οι εισαγωγέ και από τις ΗΠΑ και από τη Βραζιλία. Αντί να γίνονται αυτέ οι εκφόβιστικέ δηλώσει, γιατί δεν μπορεί να θεσπιστεί ένα σύστημα εκδηλασιμότητας. Δεν βλέπω κανένα λόγο που να είναι αντίθετο. Έχουμε ακόμα δύο θέματα, λέει ο πρόεδρο, Να ακούσουμε δηλαδή τον Πρόεδρο Γκούχτ. Ο κύριος Κάσπαρη ακόμη ζητεί το λόγο. δύο ερωτήσεις. Πρώτη, όπως του κυρίου Μάρτιν, δηλαδή το θέμα της ιχνηλασιμότητας. Εάν εν τέλει το κρέας αυτό καταλήξει στην ευρωπαϊκή αγορά, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει υποχρέωση επισήμανσης και εκεί τίθεται και το θέμα κατά πόσον είναι ανιχνεύσιμο προς τα οπίσω Ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν τεχνολογίες, τεχνολογικές δυνατότητες που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να εφαρμόσουν οι εμπορικοί μας εταίροι που να δείχνουν ότι το κρέας προέρχεται από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Και το δεύτερο ερώτημα πρόκειται για κλασική περίπτωση όπου λόγω συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δεν θα μπορέσουμε εν τέλει να αποφύγουμε την εισαγωγή του κρέατος αυτού στις αγορές μας. Ενδεχομένω να καταλήξουμε σε διαιτησία, ενδεχομένω να καταλήξουμε σε εμπορικό πόλεμο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΟΕ θα αποφασίσει κατά ε, κάθιμον. Μήπω θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε προσπάθεια να τροποποιηθούν οι κανονισμοί του ΠΟΕ να αλλάξουν οι κανόνε του ΠΟΕ ώστε να μην καταλήξει τέτοιου είδου κρέα στι αγορέ μα, Σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν κάτι τέτοιο είναι τεχνικά δυνατόν. Ωστόσο με ενδιαφέρει κυρίω απάντηση στο πρώτο ερώτημα, δηλαδή τη ιχνηλασιμότητα κατά πόσον μπορούμε να υποχρεώσουμε του ε, εμπορικού μα εταίρους να θεσπίσουν σύστημα ιχνηλασιμότητας των τροφίμων αυτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέιλορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταψηφίσει δις το κλωνοποιημένο κρέας και τώρα όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ειχνηλασιμότητας είναι δύσκολο να αποκλείσουμε ε, το κλωνοποιημένο κρέας. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι μέτρα μπορεί να, μπορείτε να κάνετε για να ε, περάσει η θέση του Κοινοβουλίου. Thank you, Ο κύριος θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο να μου διευκρινίσει κάτι, διότι άκουσα στο τέλος ότι ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει για την ε, μη εισαγωγή απογόνων, μάλλον συγγνώμη, όχι κλωνοποιημένων, αλλά απογόνων. Από ό,τι διαβάζω εγώ, είναι σχεδόν αδύνατο να έχουμε μια χνηλασιμότητα προς τα πίσω, να ξέρουμε από πού ήρθε το ζώο. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Σούλτς. Η ερώτηση μου είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Αναφερθήκατε στα κλωνοποιημένα ζώα και κατόπιν κάνατε διαχωρισμό με τους απαγόνους κλωνοποιημένων ζώων. ο Επίτροπος Ντούλη είχε πει ότι υπάρχει δυνατότητα ειχνηλασιμότητας εντός δύο μηνών. Εσείς μας λέτε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει ένα, έχετε ένα ακόμα θέμα να μας ε, αναπτύξετε πριν φύγετε. Ναι, αλλά είναι και αρκετές οι ερωτήσεις. Νομίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι θα πρέπει να κάνω τουλάχιστον μια απόπειρα να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχάς, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αλλήλως. Γιατί ακριβώς συζητάμε. Εγώ καταλαβαίνω σε εξή τη διαδικασία. Κλωνοποιούμε ένα ζώο. Αυτό που κλωνοποιούμε συνήθως είναι ένα τάβρος. Όχι αγελάδα, κλωνοποιούμε τάβρο. Ως αποτέλεσμα έχετε κλωνοποιημένους απογόνους και αυτά τα κλωνοποιημένα ζώα δεν εξάγονται. Τα κρατάτε στην κτηνοτροφική ε, σας μονάδα και αυτό που προσπαθείτε να πουλήσετε και να εξάγετε είναι το σπέρμα, όχι τα ίδια τα ζώα. Δεν θα πουλήσετε τον τάβρο, θα πουλήσετε το προϊόν του τάβρου, το σπέρμα του φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα εχνηλωσιμότητας του σπέρματος. Κατόπιν, η επόμενη γενεά, δηλαδή ε, η αγελάδα ε, λαμβάνει το σπέρμα του κλωνοποιημένου ζώου και αυτό είναι ο συνήθις τρόπος εκτροφής. Αυτό γίνεται συνήθως και με σπέρμα το οποίο προέρχεται από ταύρο ο οποίος δεν έχει κλωνοποιηθεί. Είναι η συνήθις διαδικασία εκτροφής. Και εδώ έχουμε τον απόγονο ο απόγονος λογικός δεν μπορεί να ειχνηλατηθεί γιατί είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ε, ζευγαρώματος. Και έχετε λοιπόν κρέας από απόγονο κλωνοποιημένου ζώου. Αυτά νομίζω είναι τα διάφορα στάδια. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω κατανοήσει. Αυτό που λέμε εμείς εδώ είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προ τα κλωνοποιημένα ζώα, κατανοούμε και νομίζω ότι μπορούμε και κάλλιστα να παρουσιάσουμε επιχειρήματα για την άποψή μα ενώπιον του ΠΟΕ. Τώρα, το ζώο, ο απόγονος, δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται, αλλά αν απαγορεύεται και η εισαγωγή κρέατος απογόνου, τότε ξεκινάει ένα εμπορικός, ένας εμπορικός φαύλος κύκλος διότι δεν μπορεί να ειχνηλατηθεί και καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τι γίνεται με την ειχνηλασιμότητα λοιπόν. Μπορείτε να ε, βρείτε από πού προέρχεται το κλωνοποιημένο ζώο, μπορείτε να βρείτε το σπέρμα του και εκεί σταματάει η αλυσίδα. Θα μπορούσατε ίσως να προχωρήσετε λίγο περαιτέρω και να βρείτε τον απόγονο εάν υπάρχει ένα κατάλληλο σύστημα ειχνηλασιμότητας. Αλλά ακόμα δεν διαθέτουμε τέτοιο σύστημα. Και στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει ένα εθελοντικό σύστημα ε, και μόνο δύο κτηνοτροφικά μονάδες δέχθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Ουσιαστικά λοιπόν δεν υπάρχει σύστημα ιχνηλασιμότητας. Ε, θα μπορούσε κάποιο να βάλει ένα τσίπ στο αυτί ενό ζώου, αλλά δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Τώρα, επισήμανση. Η επισήμανση ξεκινά από την προπόθεση ότι υπάρχει ειχνηλασιμότητα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε από πού προέρχεται ένα ζώο, δεν μπορείτε να έχετε και την κατάλληλη επισήμανση. Και το θέμα είναι, μπορούμε εμεί να αλλάξουμε του νόμου του ΠΟΕ. Θεωρητικώ ναι, αλλά. Ε, η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση και αυτό είναι και ένα από του λόγου για του οποίου θα αντιμετωπίσουμε πολύ περισσότερε δυσκολίε και δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάτι στην Τόχα. Ε, το να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν να αλλάξουμε μία από τις βασικές διατάξεις του ΠΟΕ είναι μία εντελώ θεωρητική συζήτηση και φαντάζομαι ότι ο κύριος Κασπαρή το γνωρίζει αυτό. Κύριε Τέιλορ, εγώ απλώς ενημερώνω την Επιτροπή σας. Στην ε, διαδικασία της συνδιαλλαγής ε, συμμετέχει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εκεί έχουμε μία διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο και το παραδοσιακό σύστημα νομοθετικής πρωτοβουλίας που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα να, να παρουσιάσει μια πρωτοβουλία δεν υπάρχει πλέον. Είμαστε στη διαδικασία λήψη απόφαση. Το Κοινοβούλιο πλέον είναι αρμόδιο να υποστηρίξει την άποψή του και δεν είναι μάλλον, δεν άπτεται τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Στάσνη, Προσπάθησα να εξηγήσω από τεχνική πλευρά τι ακριβώ εννοούμε και νομίζω ότι η τελευταία ερώτηση πάλι στην ηχνηλωσιμότητα αναφερόταν. Αυτό μπορώ να σας δώσω ως απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Ο Ντέβιτ Μάρτιν. Έχετε κάποια ερώτηση για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, αλλιώ δεν μπορώ να σα δώσω το λόγο. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Νομίζω ότι ο Επίτροπο εξήγησε πολύ καλύτερα από ότι στην εναρκτήρια του ομιλία. Εγώ νομίζω ότι η χνηλασιμότητα είναι δυνατή και υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βοηθή. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν αντίστοιχο σύστημα και δεν μπορούμε να βρούμε από πού προέρχονται τα ζώα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν είναι πρόβλημα λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πρόβλημα των ΗΠΑ και αν θέλει να πουλήσουν οι ΗΠΑ στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν ένα σύστημα χνηλασιμότητα. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Αρχίζουμε την καρτεσιανή λογική, David, τώρα. Δεν είμαστε φιλόσοφοι, είμαστε πολιτικοί και νομίζω ότι κι εσύ έχεις ένα πολιτικό βίο αντίστοιχο του δικού μου και οι ΙΠΑ δεν έχουν σύστημα εχνηλασιμότητας και δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν τέτοιο σύστημα στο εγγύς μέλλον. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να δημιουργήσουν σύστημα διότι δεν έχουν κάποια ε, ευθύνη ενώπιον του ΠΟΕ. Αυτή είναι η απάντησή μου. Θα μπορούσαν να στείλουν και τις αγελάδες του φεγγάρι αν θέλουν, αλλά δεν το κάνουν ξεκίνησαν με σκύλους, μετά πήγαν ανθρώπους. Τα πάντα είναι πιθανά σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά στον πραγματικό κόσμο, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Προχωρούμε όπως είναι τα πράγματα και αν αρχίσουμε να απαγορεύουμε την εισαγωγή ε, κρέατος από τους απογόνους θα έχουμε προβλήματα στον ΠΟΕ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Θα θέλαμε να μας πει ο Επίτροπος Δεχούχτ τι επιπτώσεις για το εμπόριο έχουμε λόγω της κατάστασης ε, στο νότιο τμήμα της Μεσογείου, κυρίως για την Τινησία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Υπάρχουν κάποια νέα ότι μπορεί να ε, ληφθούν ή έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τις εμπορικές συναλλαγές και μπορεί κατά συνέπεια να έχουμε και προβλήματα για τις δεσμεύσεις μας ως προς το εμπόριο και το εμπόριο εν γέννη στην περιοχή. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Το, αυτά που συμβαίνουν στον αραβικό, αραβικό κόσμο δεν έχουν προηγούμενο και έχουν τεράστια ιστορική σημασία. Γι' αυτό χαίρομαι που προκαλείται σήμερα συζήτηση για την εμπορική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που ε, ε, συμβαίνουν τώρα την ε, Βόρεια Αφρική. Ήδη ε, το, το Συμβούλιο τα έχει συζητήσει αυτά με πρωτοβουλία και του Πρόεδρου Βαν Ρομπόη και θα γίνει και επανεξέταση, έγκριση της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Θα μας επιτρέψει να σκεφτούμε στρατηγικά. Εάν θέλουμε το εμπόριο να συμβάλλει σε μια πιο ε, σκόπιμη, σοβαρή συνεργασία με τους Άραβες γειτονές μας θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική υπόψη μας. Όπως μπορείτε να κατανοήσετε δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να προβλέψω το ότι θα περιλαμβάνει η επικείμενη ανακοίνωσή μας. Εσείς όμως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να μας βοηθήσετε να προσφέρουμε χείρα βοηθείας στους ε, ε, Άραβες γειτονές μας. Χιλιάδες γενναίοι άνθρωποι έχουν κατέβει στους δρόμους για να διαδηλώσουν υπέρ της ελευθερίας και θαυμάζουμε το θάρρος τους. Η αφετηρία μας στο εμπόριο, ωστόσο, είναι αρκετά προηγμένη. Έχουμε ελεύθερες, ε, έχουν συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών για εμπορικά αγαθά με όλες τις χώρες περιοχής, όπως από τη Λιβύη. Στο μεταξύ έχουμε διακόψει τις ε, συζητήσεις για την Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με την Τρίπολη. Βεβαίω δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όλε οι χώρε. υπογράψαμε πέρσι συμφωνίες με τέσσερις χώρες, με το Μαρόκο. Έχουμε όμως ε, εκεί πρόβλημα ε, με την ελευθερία διακίνησης. Έχουμε τη δυνατότητα να υπογράψουμε ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. φέρνοντα οικονομίε του πιο κοντά και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω τώρα. Υπάρχει πάντοτε περιθώριο να γίνουν περισσότερα πράγματα και αν θέλουμε να παραμείνουμε σημαντικοί φορεί, σημαντικοί παίκτε στην περιοχή αυτή, πρέπει να βελτιώσουμε τι σχέσει αυτέ, εξασφαλίζοντα ταυτόχρονα ότι υποστηρίζουμε την στερέωση των ε, ε, δημοκρατικών δικαιωμάτων και της χρηστής διοίκησης. Το μήνυμα των Αράβων διαδηλωτών είναι ξεκάθαρο. Η διαφθόρα έχει σαπίσει τις κοινωνίες τους μέχρι το κόκαλο. Άρα περισσότερο εμπόριο, περισσότερες επενδύσεις θα σημάνουν περισσότερο ε, δημόσια ευθύνη. Μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα εφόσον μας ζητηθούν περισσότερα. Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως από τις χώρες μέλη και από τις δικές σας εκλογικές περιφέρειες. Δεν μιλώ κυρίως για τα δημοσιονομικά απευθύνουν έκκληση προς το μακροπρόθεσμο όραμά σας. Έχουμε υγιή σχέση, εμπορική σχέση με την περιοχή αυτού του κόσμου. 4% των εισαγωγών μας και 6% των εξαγωγών μας κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Προσφέρονται ευκαιρίες για να, βελτιώσουμε, βοηθήσουμε οικονομικά ε, μειονεκτικές κοινότητες. Ε, Άνοιγμα αγορών εκατέρωθεν της Μεσογείου πείθοντας τις κοινωνίες μας ότι δεν πρόκειται για απειλή. Πρόκειται για δρόμο διπλής κατευθύνσεως. Προσφέρει ευκαιρίες και στις δύο πλευρές. Θα προσθέσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι όταν θα διεξαγάγουμε τη συζήτηση που είπα προηγουμένω, θα μπούμε και στον πυρήνα της επιλογής αν θέλουμε ή όχι να είμαστε προστατευτικοί. Εάν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε περισσότερα υπέρ της περιοχής αυτής και νομίζω ότι αυτό πολιτικά έχει τεράστια σημασία, τότε θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να ανοίξουμε τις αγορές μας. Έχουμε προτάσεις σημαντικού εύρους που θα πρέπει πρώτα να συζητηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το σύνολο των Επιτρόπων. Θα ζητήσουμε όμως να δείξει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θάρρος για να υιοθετήσουν τέτοιες λύσεις εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί οι προτάσεις σας και αλλά και μετά τη συζήτηση αυτή κύριε Πρόεδρε είμαι διατεθειμένος να επανέλθω κοντά σας και να ξανασυζητήσουμε με λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε Επίτροπε για την ε, επίκαιρη και πολύ ουσιαστική ενημέρωση για το θέμα αυτό. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Ο Κρίστοφερ Φιέρλερ, καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν ε, σκέφτηκα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές οι οποίες θέλουν ε, να αναγεννηθούν κυρίως σε αυτό το πλαίσιο, σκέφτηκα λίγο τι κάναμε για τα Δυτικά Βαλκάνια και πώς θα απαντήσαμε στην κρίση εκεί μετά από τη δική του σύραξη. Μονομερός τους δώσαμε ελεύθερο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε μία εμπορική απάντηση έτοιμη. Είναι πολύ δύσκολο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ, διότι προσφάτως ε, με τις συζητήσεις που κάναμε συζητώντας μονομορός ε, το ελεύθερο εμπόριο ως ε, μηχανισμό υποστήριξης στην Επιτροπή μας εδώ ήταν ε, σκληρές συζητήσεις και πολύ συχνά είχαμε και αντίστοιχες σκληρές συζητήσεις στη Γενέβη. Και πάλι όμως ο επιμένων νικά και ίσως θα ήταν καλή ιδέα και σε αυτό το τομέα να προσπαθήσουμε εκ των προτέρων να ετοιμάσουμε μια πρόταση για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε και με τα Δυτικά Βαλκάνια και που προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια εξημών για το Πακιστάν. Να υπάρχει μια κάποια δυνατότητα ελευθέρου εμπορίου, ε, τουλάχιστον για την Τινησία και την Αίγυπτο. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. κύριος Κάζακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερωτησούλα κύριε Ντουχίχτ. Συζητήσαμε την τελευταία φορά Εκτός μικροφώνου ο κύριος Φιέλνερ. okay now? Okay. On avait Ο ξαναρχίζει. Συζητήσαμε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Συζητήθηκε ένα λεπτό ζήτημα όσον αφορά το αν εφαρμόζεται στην Δυτική Σαχάρα η Συμφωνία. Δεν είναι σαφές το θέμα για την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Έχει κατασταλάξει κάπου η Κομισιόν γι' αυτό. Η συμφωνία αυτή ισχύει Ιού. Ευχαριστώ, κύριε Μουσκαρντίνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ φρονώ ότι η τραγωδία που παρατηρούμε είναι κάτι που βιώνουν οι άλλοι δυστυχώς και θα πρέπει να μας οδηγήσει και στο εξής αποτέλεσμα. Εδώ και πολλά χρόνια η οικονομική πολιτική είναι στην ουσία εξωτερική πολιτική. Και εμείς εδώ και πολλά χρόνια δώσαμε βοήθεια σε κυβερνήσεις οι οποίες δεν ασχολήθηκαν με την ευημερία των συμπολιτών τους. Δικαίως λοιπόν εσείς αναφέρεστε στα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα, αλλά να είναι όμως ε, το ιδανικό ε, εμπορικό αντάλλαγμα για την βοήθεια που δίνουμε. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά θα χαθούν στον άνεμο όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να εξαγάγουμε δημοκρατία, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε ευημερία. Μπορούμε να βοηθήσουμε άλλες χώρες να βρουν τη δύναμη μέσω των λαών τους να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους σε μια πιο ισχυρή δημοκρατία και να προσφέρουμε οικονομική συνδρομή ώστε να ξεκινήσει το όλο εγχείρημα. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ το εξής. Εμείς ε, όταν συζητήσαμε για την ε, φυσική καταστροφή του Πακιστάν ε, έκτακτη βοήθεια και σε εκείνη την περίπτωση κάποιοι συνάδελφοι μέλη της Επιτροπής μας έκαναν μια πρόταση σε εσά κύριε Επίτροπο ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη σχετικά με το κατά πόσον θα μπορούσαμε να βρούμε κανόνε εντό του ΠΟΕ που θα μας διασφαλίζουν ω Ευρώπη ότι μπορούμε να παρέμβουμε εγκαίρω και για φυσικές καταστροφές αλλά και για άλλες καταστροφές που ορίστε εμφανίστηκαν. Ε, μακροπρόθεσμοι ουσιαστικά ήμασταν, διότι προβλέψαμε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν ανάλογα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε κάθε φορά να φοβόμαστε ότι θα μας μπλοκάρει ο ΠΟΕ ή να ε, ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία που ούτως ή άλλως θα μας ανακόψει την πορεία ο ΠΟΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες, κάποια κοινά κριτήρια τα οποία θα ισχύουν πάντα. Δεύτερον, σήμερα είμαστε τυχεροί διότι τουλάχιστον σε δύο από αυτές τις χώρες, έστω και προσωρινός, υπάρχει μια κυβέρνηση. Προσωρινή μεν υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά υπάρχει. Αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα ως Ευρώπη, διότι μπορούμε να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε απευθείας. Αναφέρουμε φυσικά στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση για την υποστήριξη σε επιχειρήσεις, διότι πριν γίνει πιο ελεύθερη η εξαγωγή προϊόντων και εμπορευμάτων, θα πρέπει τα εμπορεύματα να κατασκευαστούν, να δημιουργηθούν. Τι θα εξάγουν εάν η οικονομία τους ε, και η επιχειρησιακή τους ε, δραστηριότητα επιβραδυνθεί ή σταματήσει τελείως γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια θα πεθάνουν οι τοπικές επιχειρήσεις, ε, θα ε, πάψουν να υφίστανται και συμπράξεις με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ε, ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θα πωλήσουν το προσωπικό τους διότι αυτή τη στιγμή η τουριστική δραστηριότητα είναι μηδενική. Και φρονώ και με αυτό ολοκληρώνω κύριε Επίτροπε, συγγνώμη που μακρηγόρησα αλλά το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας παθιάζει εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αμέσως. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οποιαδήποτε βοήθεια αυτή τη στιγμή υπάρξει κάποια σταθερότητα και πλέον θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνει και εγγυήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις διότι η εμπορική πολιτική είναι εξωτερική πολιτική και δεν μπορούμε να την αποσυνδέουμε από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Και θα πρέπει ενώπιον του ΠΟΕ να προσπίσουμε στεναρά τα συστήματα άμεσης παρέμβασης και θα πρέπει να μην αντιτάσσετε το «ΟΠΟΕ» ε, σε εμά ε, με τους κανόνες του εμπορίου, όπως έκανε με την περίπτωση του Πακιστάν. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Κύριε Σόλτς, πρώτα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Επίτροπο για τις πληροφορίες που με τόση ειλικρίνεια μας έδωσε. Ξέρετε, την περασμένη εβδομάδα μίλησαμε με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Φίλε, he confesses that the so-called... Μας είπε και σου και μας είπε ότι υπάρχει realpolitik της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτά τα καθεστώτα και γιατί απέτυχε και αυτό διότι χρειαζόμαστε μια καινούργια, τελείως καινούργια προσέγγιση. Αυτό τονίστηκε ε, και τονίστηκε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά αυτές τις χώρες που βρίσκονται στην νότια ακτή της Μεσογείου. Τώρα, για να έρθω στο εμπορικό ζήτημα, ε, ίσως πρέπει επομένω να αναθεωρήσουμε τελείως τη σχετική πολιτική μας όσον αφορά αυτές τις χώρες. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αναθεωρήσουμε όλες αυτές τις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε και να δώσουμε την ευκαιρία σε εκείνους αλλά και σε εμάς να φροντίσουμε τα αληθή συμφέροντά μας και τα συμφέροντα δηλαδή των αντιστοίχων ε, λαών. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε η κυρία Μουσκραντίνη διότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι και το θέμα της αξιοπιστίας και το θέμα ε, του, του, του, του κύρους μας είναι σημαντικό Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα βάλουμε σε καινούργια βάση με μια τέτοια πολιτική καλή γειτονία να φροντίσουμε τι σχέσει με τι χώρε αυτέ. Επίση, κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω αν είναι δική σα αρμοδιότητα, ε, μήπω θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου μορατόριο. Μορατόριο για το εξωτερικό χρέος των χωρών αυτών διότι πηγή του χρέους είναι αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα και την ύφη πλήρωσαν οι πολίτες. Και κατά αυτόν τον τρόπο τους δίνουμε να καταλάβουν ότι τους βοηθάμε να ανασυγκροτηθούν. Φυσικά και είναι διαφορετική κατάσταση σε Αίγυπτο, διαφορετική σε Λιβύη, διαφορετική σε Τινησία. Ε, σε κάθε χώρα έχει την ιδιορυθμία της. Όμως, κατά αυτόν τον τρόπο θα τους δείξουμε ότι ε, λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση και έτσι επομένως να αντιμετωπίσουμε, να αναχαράξουμε τις ε, σχέσεις μας με αυτές τις χώρες. Ζαλεύσκη. Πάβελ Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντεχούχ που ήρθε να μας ε, πει τα θέματά του. Θέλω να σας πω το εξής. Πρώτα πρώτα θέλω να σας πω ότι όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Βορειοαφρική. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι το τέλος. Μάλλον είναι η αρχή μιας διαδικασίας. Μιας διαδικασίας που ίσως καταλήξει σε κάτι το χαόδες. Και θα πρέπει να δούμε το ότι ε, έλλειψη σταθερότητα οδηγεί στο χάος. Και μιλούμε τώρα για τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θα πρέπει να αναζητηθεί λύση. Λύση για το πώς μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, να κάνουμε δηλαδή ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε η κατάσταση αυτή να πάει προς τα εκεί που είπατε και η κυρία Μοσχαλίνη, δηλαδή να ληφθούν οι τα ανθρώπινα δικαιώματα, να γίνουν όλα όπως πρέπει για μια δημοκρατία. Τώρα, αυτή η Realpolitik σε σχέση με την, ε, τις χώρες αυτές δεν ξέρω κατά πόσο να πέτυχε ή όχι, αλλά προς το παρόν κατάσταση είναι ως εξής. Ασκούμε την πολιτική που ασκούμε ως εξωτερική πολιτική και κάνουμε ό,τι μπορούμε έχοντας επίγνωση του τι κατάσταση επικρατεί στα νότια σύνορα. Θα πρέπει όμως να βελτιώσουμε τις προτάσεις μας σε σχέση με την Λιβύη, γιατί η Λιβύη κυβερνάται τώρα από έναν δικτάτορα. Για να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε καλύτερε εξελίξεις. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι με πιο σοβαρό τρόπο να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που είπε ο κύριος Επίτροπος. Δηλαδή, Μία από τις βασικές αιτίε των εξελίξεων στις αραβικές αυτές χώρες είναι το ότι υπήρχε περιθωριοποίηση τόσα χρόνια αυτών των χωρών. Είχαμε παγκοσμιοποίηση, αλλά αυτές οι χώρες ήταν περιθωριοποιημένες και ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική κατάσταση επομένω των χωρών αυτών και τι εμπορικέ μα σχέσει να λάβουμε υπόψη όπως το τι γίνεται με την Αίγυπτο. Εξάγουμε εμεί κάτι, το παίρνουν, το αγοράζουν με κάποιοι στην Ευρώπη και μετά αυτό το εξάγουν προς την Αίγυπτο. Να ποια είναι η θέση της Αιγύπτου. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε και μια σωστή εμπορική πολιτική αλλά και επενδύσεις προς τις χώρες αυτές ούτω ώστε να προχωρήσουν τεχνολογικά οι χώρες αυτές. Αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη της οικονομίας τους. Θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσα σε αυτόν τον κόσμο της παγκοσμιοποίησης που ζούμε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητηθούν συνεργάτες, συνομιλητές που να δρομολογήσουν μια τέτοια πολιτική. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και χωρίς συνεργασία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ας πούμε, λέμε, να ανοίξει η αγορά μας προς τις χώρες αυτές. Και να προχωρήσουμε προς ε, ένα προστάδιο του ελευθερών εμπορίου. Όπως είναι σήμερα όμως τα πράγματα, δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα στην ε, Αίγυπτο, ας πούμε, δεν έχουμε ούτε ένα συνομιλητή. Πώς θα γίνουν αυτά. Θα πρέπει επίσης ότι η πολιτική χαράξουμε να είναι μακρόπνε και να είναι ρεαλιστική. Να ξέρουμε όμως τι κατάσταση επικρατεί και να βρούμε συνομιλητές της χώρας εκείνας. Πρόεδρος. Και για να κλείσουμε με αυτή τη φάση της ε, συζήτησής μας, τότε έχουμε τον τελευταίο αγορητή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. έχουμε κάποιες μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι αυτές οι μεταβολές τη κατάσταση στη Βόρεια Αφρική εν μέρη οφείλονται ή στην άνοδο των ειδών διατροφή. 2% του παγκοσμίου πληθυσμού κατοικεί στι εν λόγω χώρες. Και έχουμε 7% των δημητριακών όλο του κόσμου και 20% των εισαγωγών σιτηρών επίσης κατευθύνουν προς αυτές τις χώρες και ο πρώτος εισαγωγές στην περιοχή για το, για σιτηρά, για, για, το, στάρι είναι η Αίγυπτος. Είναι τόση ζήτηση που δεν αρκεί η παραγωγή εκεί. 20% του πληθυσμού είναι κάτω από την ηλικία των 25. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των εξαγωγών και θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο το ότι στην ε, περιοχή αυτή σε λίγο θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις εξαγωγές οπροκυπευτικών. Δεν έχουν την τεχνολογία να μπορέσουν να φροντίσουν ας πούμε το θέμα των χημικών καταλήπων. Τα χημικά στα προγυπευτικά είναι πολύ παραπάνω από τις οριακές τιμές που επιβάλλει ο νόμος. Μιλάμε τώρα για κάποιο είδου ε, λιπάσματα, ε, χημικές ουσίες που είναι απογραμμένες είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε όλο τον κόσμο. Οπότε γι' αυτό σα είπα ότι χρειάζεται τεχνική αρρωγή η Αίγυπτος και αυτέ οι χώρες. Α, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Νικόλα Ρινάλντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι οι πολίτες κάθε μέρα σχεδόν μας ρωτούν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις ε, ενδυνάμει δημοκρατίες ε, στο νότιο τμήμα τη Μεσογείου. Μέχρι τούδε η Ευρώπη δεν έχει δώσει και πολύ πιστικές απαντήσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσε ε, κάποια στοιχεία ανθρωπιστικής βοήθειας τις επόμενες ημέρες, αλλά ακόμα λείπει μια πολιτική πρόταση. Οι εμπορικές μας ε, σχέσεις από τη Συρία μέχρι το Μαρόκο είναι Συνήθω ε, μια ενιαία συμπεριφορά για όλε αυτέ τι χώρε. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή μα επιβάλλει μια διαφοροποίηση και ε, πολύ διαφορετική μάλιστα από αυτή που έχουμε σήμερα, κυρίως για να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τι χώρε οι οποίε θα ξεκινήσουν ε, μια διαδικασία εκδημοκρατισμού, εάν φυσικά προχωρήσει η όλη αυτή η διαδικασία, αλλά σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από εμά. Ο Ζαλεύσκη έχει δίκιο προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς συνδιαλεγόμενοι, αλλά μπορεί να έχουμε συνδιαλεγόμενους έξι μήνες. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε ευνοϊκές εμπορικές απαντήσεις να δώσουμε σε αυτές τις χώρες, αλλά σε έξι μήνες θα πρέπει να μπορούμε να τους δώσουμε απαντήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη χρονική συγκυρία της οργάνωσης των θεσμικών οργάνων στην Ισία και στην Αίγυπτο, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στη Λιβύη, για να προβλέψουμε κάποια μέσα εμείς άλλωστε ως ομάδα πάντα ενθαρρύναμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας πρότεινε αντίστοιχα μέτρα για το Πακιστάν. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να ε, χρησιμοποιήσουμε τα εμπορικά μέσα προκειμένου να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε σε χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Ανθρωπιστική καταστροφή στο Πακιστάν και μια νέα δημοκρατία που χρειάζεται βοήθεια σαφώς στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Θα ήθελα επίσης κύριε ε, ε, Πρόεδρε να ρωτήσω αν αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να θέσουμε μια ερώτηση στον Επίτροπο. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση για το Πακιστάν τώρα ή να περιμένω μετά. Μετά απαντω ο Πρόεδρος. Uh, let me also personally raise... Συνάδελφοι, να κάνω κι εγώ δύο ερωτήσεις. Η μία είναι επί της διαδικασίας. Από τον τύπο μάθαμε ότι η Επιτροπή είχε διακόψει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη Νομίζω ότι όλοι εδώ θα θέλαμε να είχαμε ενημερωθεί απευθεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι άλλωστε και δικαίωμα του Κοινοβουλίου κάτι τέτοιο. Η δεύτερη μου παρατήρηση. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι επί της ουσίας, διότι εδώ έχουμε τον Επίτροπο Εμπορίου και θα ήθελα να το ρωτήσω σε ποιο βαθμό μπορούμε και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά μέτρα για να βοηθήσουμε να έχουμε, ας ελπίσουμε μια δημοκρατική μετάβαση στις χώρες αυτές. Είναι στα σπάργανα η διαδικασία, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι το εφαλτήριο ενός γενικότερου εκδημοκρατισμού της περιοχής. Ελπίζουμε να είναι κάτι τέτοιο και χρειαζόμαστε μια στρατηγική, μια φιλοσοφία, να ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα πρέπει και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά μέτρα για να βοηθήσουμε τη δημοκρατική μετάβαση στις χώρες αυτές. Κατεμέ με, θα πρέπει να, να μην έχουμε ad hoc ε, ενθερμό μέτρα, θα πρέπει να επαναλάβουμε αυτό δεν μπορούμε να επαναλάβουμε συγγνώμη αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με το Πακιστάν. Θα πρέπει να έχουμε μια φιλοσοφία, μια στρατηγική, κάτι στο οποίο να μπορούμε να βασιστούμε. Το βασικό λοιπόν ερώτημα το οποίο θα μπορούσαμε να θέσουμε στον Επίτροπο Ντεχούχτ είναι κατά πόσον ετοιμάζει μια τέτοια στρατηγική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ποιο βαθμό η εμπορική πολιτική μπορεί και θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουμε την, στη δημοκρατική μετάβαση τουλάχιστον στις ε, χώρες που είναι εγκύτερες σε εμά. Μπορεί να μας ζητηθεί να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό στο εγγύς μέλλον. Το ελπίζουμε άλλωστε. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάφορα μέλη σας μίλησαν για μονομερή ενδεχόμενη εμπορική απελευθέρωση και μάλιστα για το Πακιστάν. Πρόκειται για θεομηνία, κάτι θα έπρεπε να κάνουμε δεν μπορέσαμε να το κάνουμε μέσω της ε, GSP ούτε είναι δυνατόν να το κάνουμε καθαρά μονομερός γιατί τότε πρέπει να σεβόμαστε τις σχετικές ρήτρε MFN ας το κάνουμε λοιπόν με την άρση, με το waiver συντάξαμε πρόταση, την συζητήσαμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομίζουμε ότι ήταν ουσιαστική η πρόταση αυτή αν και ήδη Είχαμε ζητήσει να μείνουν απ' έξω κάποια ευαίσθητα προϊόντα. Αλλά δεν πάνε τα πράγματα έτσι στην Γενέβη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες καταρχήν είναι αντίθετες με οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ απελευθέρωσης εμπορίου και φυσικών καταστροφών και θα είναι ακόμα περισσότερες οι αντιστάσεις αν προσπαθήσει κανείς να το συνδυάσει την απελευθέρωση εμπορίου με αναφιόμενες δημοκρατίες. Μου φαίνεται ότι θα τους φανεί πολύ πρωτοφανές το επιχείρημα αυτό στην Γενέβη. Και βέβαια τέθηκαν επιτάπητος και τα περιφερειακά στοιχεία δηλαδή των γειτονικών χωρών με το Πακιστάν εν τέλει δεν μπορούν να περάσουν οι απόψεις μας αυτές στη Γενέβη. Παρόλο που επιμείναμε πολύ, δεν περνούν οι θέσεις μας αυτές διότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Ούτε μάλιστα και με τροποποιημένες προτάσεις. Σας τα εξηγώ αυτά, αυτά για να σας δείξω τι μπορούμε θεωρητικά να φανταστούμε και τι είναι πραγματικά εφικτό στην πράξη. Ο κύριος Καζάκ Μάλιστα, μάλλον απαντώ. Λάβαμε την επιστολή του Προέδρου σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας με το Μαρόκο επί της ε, Δυτικής Σαχάρας. Αρμοδιότητα βέβαια να απαντήσει έχει κάθε άστον και θα σας απαντήσει. Η κυρία Μουσκαρντίνη ρώτησε επίσης για μονομερείς κινήσεις. Το πρόβλημα των προσωρινών κυβερνήσεων είναι βέβαια συνολικά πρόβλημα του εμπορίου. Διότι βεβαίως προϋποθέτει διαπραγματεύσεις το εμπόριο και βεβαίως χρειάζεται χρόνος πριν να μπορέσουν τα νέα συστήματα να σταθεροποιηθούν τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Ίσως μάλιστα να χρειαστεί να περάσουν και χρόνια πριν να μπορέσει να μιλήσει κανείς για μια σταθεροποιημένη κατάσταση για την ώρα. Είναι πολύ προσωρινά. Διότι η λογική της δημοκρατίας είναι ότι περιμένουμε εκλογές. Η εμπλοκή λοιπόν σε διαπραγματεύσεις με προσωρινές κυβερνήσεις δεν μπορεί να αποκλείεται αλλά θα έχει βέβαια και αυτή προσωρινό χαρακτήρα διότι μπορεί, να, μπορεί οι αποφάσεις να ανατραπούν εκ των υστέρων. Μάλιστα ορισμένε χώρες μας ζητούν να μην υποβάλουμε προσφορές σε τέτοιες ε, περιπτώσεις. Να μην ε, κάνουμε προτάσεις δηλαδή, διότι προτιμούν να τους δοθεί βοήθεια έναντι εκτιμωμένων αναγκών. Λένε για παράδειγμα ότι είμαστε εκτός δράσεως για την ώρα. Με άλλα λόγια, η πιο επίγουσα ανάγκη τους είναι επίγουσα βοήθεια εκείνη την ώρα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποκρινόμαστε, βεβαίως. Εκεί βρισκόμαστε. Ήμασταν οι πρώτοι που πήγαμε και είμαστε και πιο οργανωμένοι. Νομίζω ότι ο κύριος Σόλτς έχει δίκιο. Σόλτς, όχι Σούλτς ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις πολιτικές μας γιατί έχουμε ορισμένες, έχουμε αρκετές συμφωνίες αλλά οι παρούσες συμφωνίες δεν έχουν λάβει καθόλου υπόψη το πολιτικό σύστημα. Το έχουμε λησμονήσει εντελώ Κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις με όλους, προσπαθώντα να καταλήξουμε σε συμφωνίες, θεωρώντας ότι θα είναι υποφελή και για τα δύο μέρη. Αλλά κάποια στιγμή καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου ορισμένε χώρε πραγματικά βαδίζουν προς ένα εκδημοκρατισμό, ενώ άλλε καταλήγουν σε απόλυτη αστάθεια. Και βεβαίω έχουμε και όλε τι ενδεχόμενες περιπτώσεις ενδιαμέσως Για το χρέος προτιμώ να μην εκφραστώ διότι δεν έχω και ιδέα ποια είναι η χρέωση των χωρών αυτών. Ίσως να μην απαραίτητα τόσο υψηλά τα χρέη τους. Είναι πάντως κάτι όπου δεν μπορώ να ε, εκτιμήσω. Ο κ. Ζαλεύσκη σωστά μίλησε για το πρόβλημα του συνομιλητού. Βεβαίως πρώτα πρέπει να βρούμε συνομιλητή. Βέβαια οι τιμές των τροφίμων παίζουν σημαντικό ρόλο και συζητούμε για την ώρα με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστότερα το θέμα. Το συζητούμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Ρινάλντι. Κυρία Ρινάλντι, νομίζω ότι χρειάζεται ναι, νέα κύριος Ρινάλτη, συγγνώμη, ε, κατηγορία αναφιόμενων δημοκρατιών, αυτό πρέπει να ζητηθεί στην Γενέβη και άλλοι βουλευτές το έθεσαν. Το θέμα έχει πολιτικό χαρακτήρα. Βέβαια, στη Γενέβη η συζήτηση είναι καθαρά εμπορική. Και σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή ισχύω των συμφωνιών, οι διαπραγματεύσεις οι για συμφωνία με τη Λιβύη είχαν μεικτό χαρακτήρα και εμπορικό και για άλλα θέματα. Η κυρία Άστον δήλωσε ότι έχουν ανασταλεί οι διαπραγματεύσεις. Εγώ συμφωνώ βεβαίω, ε, ε, ασφαλώς με αυτό. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και να διαπραγματεύεται υπό τις συνθήκες αυτές. Κατανοώ βεβαίω την απάντησή της και σε μένα να είχατε θέσει την ίδια ερώτηση θα είχα απαντήσει το ίδιο πράγμα και χωρίς περαιτέρω διαβουλεύσεις με κανένα. Είναι, είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται διαβούλευση με κανένα πριν να το πείτε αυτό. Αναστολή των διαπραγματεύσεων είναι και απλή όταν είστε μέρος των διαπραγματεύσεων. Δεν ξαναπάτε. Αυτομάτως αναστέλλονται δεν είναι θέμα να υπάρξει απόφαση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εάν δεν διαπραγματεύεστε πλέον, αυτομάτως, de facto, αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις. Προσπάθησα, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στις περισσότερες τουλάχιστον ερωτήσεις. Μήπως λησμόνησα καμία. Σας ευχαριστώ. Νικολάρη, νομίζω ότι καλυφθήκατε για το Πακιστάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα με το Πακιστάν είναι το ότι, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι το ότι δεν έχει σημειωθεί στη Γενέβη ε, πρόοδος στις συνομιλίες. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το κατά πόσο θεωρεί η Κομισιόν ότι αν εμεί κάνουμε μια ψηφοφορία αν, επί κάποιο κειμένου, αν αυτό θα βοηθήσει τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στη Γενέβη. Ή θα πέσει το κενό ο κ. Επιτρόπος. Το Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο να αποφασίσει ότι θέλει να θα κάνει κάτι τέτοιο. Προσωπική μου άποψη πάντω είναι ότι δεν πρόκειται η διαδικασία τη Γενέβη, οι συνομιλίε να ωφεληθούν. Ίσως ε, δείξουμε και κάποια ετοπάθεια. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι οι πρωταγωνιστές του έργου δεν θέλουν να προχωρήσουν, να απεμπλέξουν το θέμα. Πάντω, αν θέλει το κοινοβούλιο να ψηφίσει, α ψηφίσει το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πιτροπολίτη, Πρόεδρο. Επομένω, το ολοκληρώνουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντεχιούχτ που ήρθε να μα ενημερώσει. Και μα ε, απάντησε σε αυτά τα θέματα. Τώρα, ζητώ να με καταστήσει αν θέλει ο Παύλ Ζαλεύσκη για λίγο ε, μέχρι ότου ξεβγάλω μέχρι την έξοδο συνοδεύσω τον κύριο Ντεχούχτου. Ladies and gentlemen, I would like to proceed further. Uh, we have some points uh, to the end of our... Συνεχίζουμε Σε εργασίες επιτροπής μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο θέμα είναι το υπερμαριθμό 10. For a post-crisis world. Uh. Η προσαρμογή της Ευρώπης με μια ένωση καινοτομία για ένα κόσμο μετά την κρίση. Η Νέζ Βάιντερ που είναι η συγγήτρια δεν μπόρεσε να προσέλθει αλλά ο κύριος Κάσπαρη έχει ασχοληθεί με την έκθεση ε, και υποβάλλει τροπολογίες. Οπότε μπορεί να μας διαφωτίσει ο κύριος Κασπάρη. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος η συνάδελφος μάλλον ε, λείπει γιατί συμμετέχει σε άλλη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα διαβάσω λοιπόν τα όσα μου γράφει. Μου λέει λοιπόν, εάν εγνώριζα ότι θα συμπέσει με το ίντα θα είχα ακυρώσει την συμμετοχή μου. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν, δεν ήταν πλέον δυνατό. Σας ευχαριστώ για τις σημαντικές συνεισφορές σας στην εργασία μου. για σημαντικά θέματα όπως τις, ε, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, θέματα δηλαδή που χρειάζονται μελέτη, μέχρι και για θέματα ε, δημοσίων προμηθειών πέραν των συνόρων. Έχω εξετάσει τα τις σχετικές τροπολογίες προσεκτικά. Ευχαρίστως θα περιλάβω την μεγαλύτερη ε, το μεγαλύτερό τους αριθμό στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Η γνωμοδότηση θα αναφέρει ότι πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και περιβαλλοντικές σκέψεις να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτάρκεια σε ενέργεια, να προστατεύονται ε, η πνευματική διοκτησία και τα άλλα από ε, κατάλληλες διατάξεις. Όλα αυτά πρέπει να υποστηριχθούν. Επίσης, βρήκα σημαντικό συμπλήρωμα του αρχικού κειμένου του σχεδίου γνωμοδίσεως τις τροπολογίες που ζητούν ενισχυμένη υποστήριξη και στα πλαίσια των στατικών στόχων της Ευρώπης 2020, η ανάγκη αντιμετώπισης μη δικαιολογημένων εμπορικών ε, φραγμών και ούτω καθεξής. Ορισμένες τροπολογίες δεν μου φάνηκαν συμβατές, θα χρειαστεί να γίνουν ορισμένες συμβαστικές τροπολογίες, θα τις υποβάλω σε όλους τους ενδιαφερομένους. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να έρθετε σε επαφή μαζί μου αν έχετε παρατηρήσεις να μου υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τα λόγια της συναδέλφου μου και ευχαρίστω να μεταφέρω όποιους απόψεις εκφραστούν εδώ. Thank uh, Now it's time. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να βγουν τον λόγο τα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Άντερ, Άντερ θα μιλήσω εγώ εκ μέρους του εισηγητού κ. Μπαλσάνι, που είναι συντάκτης ε, και ε, μου είπε, δι' αυτό το σημείο, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ε, το, το έργο του, να τον ευχαριστήσω επίση για το ότι δέχεται του συμβασμού, για, για τη συνεργασία και θα πρέπει να σα πω ότι στο, πάρκο, στο πλαίσιο αυτών των ε, πολιτικών καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερω τα εξή. Πρώτα-πρώτα, να βοηθήσουμε την παραγωγή και την τεχνολογία που είναι συμβατή με το περιβάλλον και θα πρέπει να έχουμε οικονομία σε ενέργεια, όχι πολλές εκπομπές διοξιδίου και να προστατευτεί η πνευματική διοκτησία. Να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να γίνει χρηματοδότηση και να γίνει εσωτερήκευση των, των δαπανών, να σταθεροποιήσουμε τα επιτόκια, να υπάρξει περισσότερη προστασία νομική ε, των επιχειρήσεων ως προς τις άλλες χώρες και να, προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας από τις παραποιήσεις και απομιμήσεις και επομένως θα πρέπει να κάνουμε αυτή την πολιτική καινοτομία σε ένα όχημα, ένα μέσο για απασχόληση, να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη παντού για την στρατηγική για το 2020 και γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανταγωνιστική εμπορική πολιτική και αυτό είναι βασικό για να μπορέσουμε να φτάσουμε το 3% της 100 που θέλουμε όσον αφορά την, την ανάπτυξη και θεωρούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα έρευνα, να το χρηματοδοτήσουμε για να έχουμε περισσότερη, περισσότερη ανταλλαγή ε, σε διεθνές επίπεδο για τις εμπορικές ε, συναλλαγές και να βοηθήσουμε για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Ό,τι θέλετε πέστε μου και εγώ το διαβιβάσω στον εισηγητή. Πρόεδρε. Εγώ θα πω για την εξήγηση του κύριου Τζενάρο που δεν είναι σήμερα εδώ. Έχει κατεβάσει εννέα τροπολογίε για την εν λόγω έκθεση. Και ελπίζει ότι κάτι θα προσθεθεί στην ε, έκθεση αυτή. Θα πρέπει να βλέπουμε πιο συγκεκριμένα λέει, για το τι θα κάνουμε, πώς θα μετασχηματίσουμε την Ευρώπη σε αυτόν τον κόσμο μετά την κρίση. Παρακαλούμε και οι άλλες πολιτικές ομάδες επίσης να δείξουν κατανόηση, να συμφωνήσουν και έτσι να έχουμε μια επιλεκτική εσωτερήκευση και κάθε τον τρόπο να έχουμε μια αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική και στρατηγική. Να προσέξουμε τους τομείς πραγωγής όπου μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικό συγκριτικό πλεονέκτημα την επόμενη 20 και επίση να κάνουμε μια στροφή όσον αφορά κάποιε φιλικέ προ το περιβάλλον, προ την αλλαγή του κλίματο και αποτελεσματικέ ε, δομέ στην ε, βιομηχανία, να προσέξουμε να καλύψουμε την εσωτερική ζήτηση, διότι νομίζουμε ότι η εσωτερήκευση να είναι κάτι σαν προσθήκη και όχι υποκατάστατο για να έχουμε μια υυξημένη εσωτερική ζήτηση. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίσουμε καλύτερα τους αδικαιολόγητους δασμολογικούς φραγμούς. Καλύτερη νομική προστασία να γίνει και να υπάρξει περισσότερη διάδοση της τεχνολογίας παντού. Ευχαριστούμε κύριε Τελεόρ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Um, Daniel, Mr. Kaspari, you would like to comment το λόγο. Όχι, όχι, ο κ. Κασπάρη. Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να σχολιάσει. Όχι. I Για να δούμε τι, τι προθεσμίες έχουμε. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στη συνεδρία της 15ης ή 16ης Μαρτίου. That is uh, uh, the voting in the committee. Now we Τότε, τότε θα γίνει ψηφοφορία ή στην Επιτροπή. Και τώρα προχωρούμε. Πάμε στο σημείο παριθμών 11. Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Έκθεση Σλίτερ Δεν είναι όμω εδώ. Και πάμε στο επόμενο. Μπα και εντωμεταξύ έρθει ο κ. Σλίτερ. Uh, this Οπότε θα ξαναγυρίσουμε στο 11. Πάμε επομένω στο 12 η Ευρωπαϊκή Ένωση ω παγκόσμιο φορέα και ο ρόλο τη στι πολυμερεί οργανώσει. Έχουμε τώρα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία τη ΑΦΕΤ για τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης πολυμερεί οργανώσει. ξαναλέει ο πρόεδρο. Οπότε θα πρέπει να διερευνήσουμε τι δυνατότητε παρέχει η συνθήκη τη Λισαβόνα, ώστε να προβάλλεται η Ένωση έτσι που να μπορεί με μία φωνή να τοποθετείτε, να εκπροσωπείτε εις το διεθνή στίβο. Ο κύριος Λάιχτφριντ από τους σοσιαλιστές και Δημοκράτε θα πρέπει να λάβει το λόγο. Αλλά στη θέση του θα μιλήσει ο κύριος Μάρτιν. Mr. So, Mr. Martin, please, the floor is yours. Έχετε το λόγο κύριε Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ επί τη βάση σημειώσεων που μου έδωσε ο Γιώργ. E Συζητάμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμια φορέα στις πολυμερές οργανώσεις και εξετάζουμε τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να μιλά με μία φωνή σε διεθνή φόρα. Η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, έχει και κάποιες συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο φορέα για τις πολυμερείς ε, οργανώσεις ε, στο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα της παγκόσμιας διακυβέρνηση και στις ομάδες G, G8, G20 κτλ. και τις σχέσεις τους με το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας ενδιαφέρει και απάντηση στη σχέση με τον ΠΟΕ ο ΣΥΝΤΑ και η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, κατόπιν συμφωνίας δεν θα περιλαμβάνει σχόλια επί του θέματος, θα, θα βασιστεί στη δική μας γνωμοδότηση. Ε, θα αναφερθούμε λοιπόν από πλευρά μα στον ΠΟΕ και ίσω αργότερα θα μπορέσουμε να καταθέσουμε και τροπολογίε για άλλου οικονομικού οργανισμού. Ιστορικός η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νομικός και πολιτικός ε, δεσμευμένη για την ε, πολυμορφία της που είναι ο βασικός τρόπος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξωτερικά θέματα. Ε, το συστήματά μας μας παρέχουν νομική σαφάνεια, ε, σαφήνεια και διαφάνεια και είναι ένα πολύτιμο μέσο για να έχουμε ε, καταλληλότερη διαχείριση με πιο πειθαρχημένο τρόπο και να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες μέλος του ΠΟΕ συμμετείχε στις δομές οι οποίες είναι υπεύθυνε ε, για το παγκόσμιο εμπόριο, όπως για παράδειγμα τη συζήτηση που είχαμε το 1995 στον ΠΟΕ και επίσης συμμετέχουμε στο παγκόσμιο εμπόριο μέσω και της δικής μας ε, εμπορικής πολιτικής. Η επέκταση της ε, Εμπορική πολιτικής που καθορίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα, που περιλαμβάνει πλέον και τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις δίνει μια πιο ισχυρή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντό του ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά μπλοκ, που σημαίνει ότι είναι ένα από του βασικού παράγοντε στον ΠΟΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά με μία φωνή. Ο Επίτροπος Εμπορίου είναι αυτό ο οποίο διαπραγματεύεται εξ ονόματο όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στον ΠΟΕ ανεξάρτητα, αλλά συμμετέχουμε και ω ενιαίο μπλοκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει επίση. Αντίστοιχα, ε, αντίστοιχη συμπεριφορά δεν έχουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενέβη από το 2011 και μετά έχει δύο αντιπροσωπείες. Τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΠΟΕ και τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών φορέων στη Γενέβη. Το σκεπτικό είναι να υπάρχει σαφή καταμερισμό εργασία και να μπορεί να διευκολυνθεί το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ενίσχυση τη παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διάφορε οργανώσει που εδρεύουν στη Γενέβη. Περιλαμβάνεται και μια κοινωνική πτυχή για το εργασιακό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία μπορεί να έχει σημαντικέ επιπτώσει ε, για την αλλαγή των ε, μελών του ΠΟΕ και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε και να αναλάβουμε και τι ανάλογε ευθύνε θα πρέπει να σεβόμαστε τις εμπορικές εμφανίες ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι δραστήρια και να ενισχύσει το ρόλο της Γενικής Γραμματείας του ΠΟΕ, να παρέχει τεχνική συνδρομή, κυρίως στα μέλη του ΠΟΕ. Ο ρόλος της Γραμματείας του ΠΟΕ είναι πολύ σημαντικός και Γι' αυτό λοιπόν είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει εκπροσώπηση αξιωματούχων από ανεπτυγμένε και αναπτυσσόμενες χώρες για να είναι ο ρόλος αυτό πιο αποτελεσματικό. Όσον αφορά τώρα την αρχή της συνένεση στη διαδικασία λήψη αποφάσεων του ΠΟΕ, εξετάζουμε ακόμα εναλλακτικέ λύσεις προκειμένου να διευκολύνουμε μία αναπερίπτωση εξέταση του κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε συνένεση. Το να καθορίσουμε καλύτερα τις δραστηριότητες και τους νέους κανόνες οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή υφιστάμενων συμφωνιών ε, είναι εξίσου σημαντικό και μας ενδιαφέρει επίσης να υπάρχει διαφάνεια στις εμπορικές πολιτικές ε, και αυτή είναι μία εκ των όνου κάνευ ε, απέτηση των πολιτών του κόσμου. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί η δράση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή των υποχρεώσεων του ΠΟΕ και η αξιοπιστία του συστήματος επίλυση διαφορών μπορεί ε, να εφαρμόζεται και με πρακτικό τρόπο βάσει των συστάσεων του ΠΟΗ και στα πλαίσια του ΠΟΗ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει συνέπεια της εμπορικής πολιτικής με άλλες ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως την ανάπτυξη και θα πρέπει να έχει έναν ηγετικό ρόλο στον ΠΟΕ, ώστε οι δράσει που αναλαμβάνει να είναι αντίστοιχε με τις δράσεις ε, που αναλαμβάνουν άλλε οργανώσεις. Όπως σας είπα, αυτές είναι οι συστάσεις του Γιώργ. Εγώ τις διάβασα για πρώτη φορά και συμφωνώ, αν όχι με, τις ε, αν όχι με όλες, με τις περισσότερες από αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιο να μιλήσει από τα μέλη. Κύριε Σότ. ευχαριστώ. Και εγώ μόλις άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την εισαγωγή του συναδέλφου για την ε, προσέγγιση που ακολουθεί όλη η γνωμοδότηση και νομίζω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στα, θέματα του ΠΟΕ όπως μόλις συζητήσαμε με τον Επίτροπο. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να κάνουμε μια πιο διεξοδική ανάλυση και να παρουσιάσουμε πιο αναλυτικές απόψεις για το ρόλο μας ε, στους διεθνείς οργανισμούς ε, σε θέματα εμπορίου. Είμαι καθόλου διαθέσιμος να συνεργαστώ με τον συντάκτη της γνωμοδότησης ως ε, σκιώδη συντάκτη. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Άλλος, κανείς. Όχι. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποτελεσματικότητά της. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Because... Ουδής. Λυπάμαι, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συζητήσεις μας. Θα μας ενδιέφερε πολύ να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Σήμερα γίνεται μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κατόπιν θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης στις 15 Μαρτίου μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η οποία γίνεται σήμερα, παρεπιπτόντω. Κατόπιν, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης. Μάλλον, στις 22 Μαρτίου. Και η ψηφοφορία της γνωμοδότησής μας στην Επιτροπή 13 Απριλίου. Κατόπιν, η εξωτερικών υποθέσεων θα, θα ψηφίσει συγγνώμη, στις 20 Απριλίου για την έκθεσή της και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαΐου. Ο κύριος Σλίτερ είναι πλέον αίθουσα. επομένως μπορούμε να επανέλθουμε στο σημείο 11. Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. εισηγητής ο Καρλ Σλίτερ και σήμερα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Πρόκειται για τη δεύτερη εξέταση των τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης για την ε, πρόταση του συγκεκριμένου κανονισμού. Προθεσμία για τις τροπολογίες ήταν η 20 Ιανουαρίου. Ε, 184 ε, τροπολογίες στο σύνολο. Εχθές ε, διοργάνωσε μια συνάντηση ο κύριος Σλίτερ επί του θέματος. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κάποια τεχνικά προβλήματα στο τηλεοπτικό στούντιο είχαμε. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το πόσο προκάλεσε την προσοχή του κόσμου το θέμα αυτό. Οι επενδύσεις από την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλες και οι επενδύσεις στην Ευρώπη αυξάνονται και κάποιες από αυτές τις ε, συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές για τις επιχειρήσεις ε, που επενδύουν. Και ο κόσμος ε, φοβάται πολύ για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι συμφωνίες. Αλλά διαπίστωσα ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θέλουν να γίνει αυτή η μετάβαση με λογικό και κατάλληλο τρόπο. Συνεπώς, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε και ε, συμβιβασμούς με τους οποίους θα μπορούσαν να συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, εάν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε επιρροή στο Συμβούλιο, να συμφωνήσουμε εμείς τουλάχιστον εδώ, θα πρέπει να δεχτούμε βέβαια ότι τα πάντα δεν είναι ρόδινα. Και όπως και να έχει, το Συμβούλιο δεν πρόκειται να δεχτεί την ε, πρότασή μας απαράλλαχτη. Εάν λοιπόν δεχτούμε όλοι ότι αυτό είναι το προϊόν που δώσαμε για διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε από αυτού και κατόπιν να δούμε πόσο ε, βαρύτητα έχει το Συμβούλιο, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Αν δεν συμφωνήσουμε από αυτού, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη μακρά οδό. Ε, το Συμβούλιο προς το παρόν δεν μας έχει δώσει καμία ένδειξη γιατί περιμένουν εμά. Από όλε τι τροπολογίε διαπίστωσα ότι οδεύουμε προ όλε τι κατευθύνσει. Και Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία είναι εν εξελίξη και μεταξύ ημών και μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Ε, οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ μου είπαν τι προσπάθειες κάνετε εσείς να καταλήξετε σε κάτι. Κάναμε και μια συνεδρίαση εχθές με τους κοιόδης εισηγητές για να δούμε πού υπήρχε περιθώριο να έχουμε κάποιο σημείο επαφής. Σήμερα ε, μάλλον να πω ότι πρώτον ε, ήρθα σε επαφή με κάποια από τα μέλη που κατέθεσαν τροπολογίε. τι δυνατότητες έχουμε για συμβιβασμούς. Μετά από αυτές, ε, αυτή τη συζήτηση θα κάνω κάποιες προσαρμογές στις περισσότερε από τι τροπολογίε. Ελπίζω να τι έχω έτοιμες το απόψε, αλλά αύριο το πρωί μάλλον θα τι στείλω και να δούμε τι περιθώριο κινήσεων έχουμε. Τα περιθώρια που έχουμε είναι τα εξής εμείς συμφωνούμε όλοι, νομίζω, ότι κάποια από τα παλιά στοιχεία θα παραμείνουν. Η προϋπόθεση είναι να μην ε, υπάρχουν προβλήματα με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί και πέρα οι χώρες μέλη μπορούν να κάνουν νέες συμφωνίες, αλλά και πάλι συμφωνούμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι οι συμφωνίε αυτές δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη νέων μελλοντικών ευρωπαϊκών συμφωνίων. Όταν μια χώρα ξεκινά και θέλει να κάνει μια νέα συμφωνία, θα πρέπει να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκή συμφωνία. Ως προς αυτό φαίνεται ότι συμφωνούμε. Τώρα, το πότε έχει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναδιαμα πρευτεί ή να ζητήσει να επαναδιαπραγματευτεί ή να αποσύρει την πρότασή τη, φαίνεται ότι διαφωνούμε. Σε αυτό που συμφωνούμε όλοι είναι ότι όπου υπάρχει αντίφαση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τότε ε, συμφωνούμε όλοι επί του θέματος. Οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε επίση συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις πολιτικές, πρέπει να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση, αλλά αν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική, διαδραματίζεται κάποιος ρόλος ε, της πολιτικής αυτής. Η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα νωρίτερα ήταν σαφής ότι πρέπει να έχουμε ένα συνδυασμό πολιτικών και εμπορίου. Εδώ φαίνεται ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει τουλάχιστον να παρακολεί τις πολιτικές που είναι γραμμένες στη συνθήκη. Νομίζω ότι εδώ είναι το σημείο στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Επίσης, συμφωνήσαμε όλοι ότι η διαφάνεια δεν είναι το πώς θα το αντιμετωπίσουμε και σε ποια άρθρα ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει, αλλά η διαφάνεια είναι σημαντική και επειδή πλέον η αρμοδιότητα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε κάποια σημεία φαίνεται ότι θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχει διαφορά. Όταν υπάρχει θέμα επίλυσης διαφοράς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τουλάχιστον πρόσβαση. Σήμερα μπορούν αλλά δεν έχουν πρόσβαση στην ε, τεκμηρίωση. Οι περισσότεροι από εμά δεν καταλαβαίνουν πού είναι η λογική σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάγιε σταθερέ διαδικασίε για την ε, εμπιστευτικότητα, αλλά δεν του επιτρέπεται να δουν ούτε τα έγγραφα. Οι περισσότεροι εξημών θεωρούμε ότι κάπου υπάρχει ένα λάθο αυτό όλο. Νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση ήταν ε, αρκετά καρποφόρα και ευχαριστώ όλες τις ομάδες γιατί ναι μεν ήταν δύσκολη συζήτηση αλλά προχωράμε με αργά βήματα προς μια κατεύθυνση. Νομίζω ότι κοντεύουμε να συμφωνήσουμε αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία για άλλη μια ε, συνεδρίαση ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινά σημεία επαφής γιατί αυτό θα διευκολύνει τη συζήτησή μας με το Συμβούλιο. Ε, έχω την ε, αίσθηση ότι πλησιάζουμε, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποιον επιπλέον χρόνο για να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, θέλουμε να έχουμε επενδύσει και να προχωρήσουν και τα άλλα μα συμφέροντα καταλήλω και να αντιλαμβάνονται όλο το κείμενο με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να ετοιμάσουμε ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο και αυτό φυσικά θα διευκολύνει και τι εργασίε μα με το Συμβούλιο και να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μα αργότερα. Με αυτά νομίζω ότι ολοκλήρωσε την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Ως και ο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας, για αυτό που προσπαθήσετε να κάνετε για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εξημών ε, εκτιμούμε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Τα μέλη τώρα. Ο κύριος Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα των επενδύσεων και το τι κάνουμε με τις διάφορες υφιστάμενες συμφωνίες δικαίως μας απασχολεί και τόσο εντατικά και ευχαριστώ τον εισηγητή που αφιερώνει και πολύ χρόνο στις συνομιλίες με τους κοιόδης εισηγητές αλλά και άλλους συναδέλφους και θα, προσπαθήσουμε να, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ορθή λύση. Το δικό μου πρόβλημα και εγώ ακόμα αμφιταλαντεύομαι είναι η παράγραφοι 5 και 6. Τι θα κάνουμε με τις υφιστάμενες συμφωνίες. Κάτι που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μάλιστα το έχω επαναλάβει αυτό εδώ στην παρούσα Επιτροπή, η Επιτροπή λοιπόν έχει υπνώσει επί σειράν ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για τις διμερείς συμφωνίες προστασίας, αλλά θεματοφύλακας των συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ λοιπόν θεωρώ Έχω δυσκολία να πιστέψω ότι όλες οι υφιστάμενες ε, συμφωνίες προστασίας τίθενται υπό αμφισβήτηση. Βλέπω όμως με κάθε μέρα που περνά εδώ στο Κοινοβούλιο και που συζητούμε για τις υφιστάμενες συμφωνίες βλέπουμε την κατάσταση στις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τις συμφωνίες αυτής τη προστασίας. Οι επιχειρήσεις βλέπω να γίνονται πιο νευρικές καθώς επίσης και οι εταίροι μας στο εξωτερικό και κυβερνήσεις και επιχειρήσεις παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συζητήσεις και με ιδιαίτερη ανησυχία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ναι μεν συμφωνούμε σε πολλά θέματα εδώ, παρόλα αυτά θα πρέπει όλοι να καθίσουμε να σκεφτούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των τρέχουσών συζητήσεών μας, ιδίω για τις παραγράφους ή άρθρα 5 και 6, ποιες είναι οι επιπτώσεις στους εταίρους μας αλλά και στις επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πράγματι πώς παρόλες τις, παρόλες τους αγώνες που θα κάνουμε για τις μελλοντικέ συμφωνίες προστασίας και θα βρούμε βεβαίως κάποια σημεία που θα συμφωνήσουμε θα πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε να επιφέρουμε κάποιες ζημίες. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον εισηγητή για τον χρόνο που αφιερώνει και είμαι και αισιόδοξο πράγματι ότι θα βρούμε λύση, αλλά παρακαλώ και πάλι να σκεφτούμε προσεκτικά ποιε είναι οι επιπτώσει των ενεργειών μα στι επενδύσει παγκοσμίω. Thank Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Κασπέρο, Φιέλνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα όσα λέει ο Καρλ Σλούτερ ηχούν θετικά σχετικά με την εξέβρεση κοινού εδάφους. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, λέει ο κύριος Χέλνερ. Πάντως, όπως είπε και ο προλαλής σας Ντάνιελ Κάσπαρη, θεωρώ ότι τα πιο ευαίσθητα σημεία είναι η παράγραφη η 5 και 6 και πώς θα διασφαλίσουμε ε, ασφάλεια δικαίου. Βρίσκω λίγο δύσκολο να είναι δυνατόν να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τις υφιστάμενες συμφωνίες, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τις αποσύρει νομίζω ότι ε, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί τεχνική λύση για να υπάρξει μια κατάλληλη ισορροπία, διότι πραγματικά πρόκειται περί ακροβασίας ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες. Αφενός λοιπόν οι υφιστάμενες συμφωνίες που πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται και ταυτόχρονα θέλουμε να δώσουμε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποχωρεί από συμφωνίες που θεωρεί ότι είναι ανεπιθύμητες για κάποιο λόγο. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου. Ένα άλλο πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει είναι το δικαίωμα της Κομισιόν να διορθώνει σφάλματα χωρίς να εμπλέκεται το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή χωρίς μέλη. Διαρωτώ με αν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα, θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει μέσα σε ένα έτος τις πέντε περίπου χιλιάδες ε, υφιστάμενες συμφωνίες. Πάλι εδώ βλέπω λοιπόν να μην υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Η Κομισιόν είναι θαυμάσιο θεσμικό όργανο, αλλά πώς θα τα καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα έτος δηλαδή, να βρει τα σφάλματα 5.000 συμφωνιών. Εγώ βρίσκω ότι αυτά δεν είναι ρεαλιστικά. Πρέπει να βρούμε κάποια διαφορετική και πιο πρακτική λύση. Αυτά είναι πάντως τα, τα, θέματα που, που ε, ε, ε, προσήλξαν την προσοχή μου. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα διμερώς για να εξετάσουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά αυτά είναι τα βασικά θέματα που ήθελα να θέσω τώρα και ελπίζω επαναλαμβάνω να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση που να προσφέρει ασφάλεια δικαίου. Σας ευχαριστώ Χρήστοφερ. Άλλος κανείς που επιθυμεί να εγείρει την φωνή του επί του προκειμένου θέματος. Ίσως τότε εγώ ως Κιώδης να μιλήσω και από πλευράς του ΕΛΚ να σας πούμε τη θέση μας θεωρώ ότι έχει διαμορφωθεί μια συνένεση αυτό είναι αδιαμφισβήτητο όλοι συμφωνούμε το θέμα δηλαδή του πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο μέλλον για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά αυτές τις ας τις πούμε επενδυτικές συμφωνίες Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει, να αναλάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και θα πρέπει να έχει την καταλή εντολή. Πολύ θετικά είναι τα πράγματα, μια που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι εκ των εταίρων μας θα ήθελαν να αναλάβει αυτόν τον ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ βασικό. Για να είμαστε ρεαλιστές πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι διμερείς ισχύουσες συνθήκες. Υπάρχει πάντως για αυτό τον τομέα περιθώριο συμβασμών. Και άρα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι σχετικές απόψεις. Ε, να σας πούμε τη θέση του ΕΛΚ. Τι θα γίνει δηλαδή όταν οι σημερινές επενδυτικές ε, ούτως συμφωνίες τεθούν ένα αμφιβόλο. Έχουμε το άρθρο 21 τη συνθήκη που προβλέπει πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι δυνατόν να συνεχίσουν να ισχύουν αυτέ οι συμφωνίε και με αυτόν τον τρόπο πάβει να υπάρχει ασφαλεία δικαίου. Αυτό ακριβώ που ετώνησε ο κ. Κάσπαρη ότι πρέπει να ισχύει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό θέμα στο μέλλον. Όλοι θέλουμε να έχουμε τέτοιες συνθήκες. Θέλουμε να υπάρχει κοινή επενδυτική πολιτική που όμως να ε, είναι σε ένα πλαίσιο άρτιο νομοθετικό. Και ακούγοντας και την γνώμη του κύριου Κάσπαρη θα πρέπει να πούμε και εμείς ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σχολιάσουμε για το τι θα γίνει με αυτές τις συμφωνίες στο μέλλον. Και πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ σύντομα προς την κατεύθυνση αυτή της υιοθέτησης δηλαδή μιας θέσης. Και όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο στι επαφέ και διαπραγματεύσει με του ε, διεθνεί συνομιλητέ μα. Πάντως πρέπει και πάλι να συγχωρούμε τον κύριο Σλίτερ, ο οποίος έκανε την μπορούσε για να επιτευχθεί συμβιβασμό. Έχει το, το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Κρίστοφερ, Ντάνιελ, είναι σαφέ αυτό το οποίο είπες, ότι το άρθρο 5 και άρθρο 6 είναι το πιο σημαντικά όσον αφορά την ισχύουσα συμφωνία. Δηλαδή είναι η αναθεώρηση της ισχύουσης συμφωνίας και οι συνέπειες αυτής ή των ισχυουσών συμφωνιών. Τα τρία τρίτα της μας αφορούσαν, όταν βρέθηκα με τους άλλους σκιώδες, αφορούσαν ακριβώς τα σημεία αυτά. Καμιά φορά δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο στεγανό 100% σύστημα και άλλωστε κανείς δεν το θέλει ενδεχομένω γιατί δεν είναι δυνατόν να θωρακίσουμε 100% καμία πολιτική. in achieving the policies of the Union and define them very nicely. That is not even... Αυτές οι ρήτρες, οι δεόμενες sunset καταληκτικές, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. μη φοβάται συμφάστε στην εμπορική πολιτική δεν μπορεί να μπει δικτατορία. Πάντως έχει διαμορφωθεί μια πλειοψηφία. που θεωρεί ότι μπορεί να στεγανοποιήσουμε την κατάσταση. Μην δημιουργήσουμε όμως και αδικαιολόγητους φόβους ούτε κάποιες, κάποια πολιτική επενδύσεων που είναι τελείως άσχετη με τις άλλες πολιτικές. Να υπάρξει κάποιο είδους ασφάλεια για τις επενδύσεις και γι' αυτό και θα πρέπει να ξαναπούμε ότι πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα με κρατικά μονοπόλια από κάποιων χωρών σε σχέση με τα χρήματα που θέλουμε να επενδύσουμε που είναι αρκετά δεν είναι δυνατόν επομένω να απομονωθεί, να αποστασιοποιηθεί αυτή η πολιτική. Ήδη έχουμε το άρθρο 258 τη συνθήκη, όπως είπε και ο κύριος Φιέλνερ. Ε, είπαμε ότι έχουμε τώρα το θέμα ένδικης επίλυση διαφοράς. Άρα, θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουμε προς εξέβρεση λύσεως. και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι τόσο προβληματισμένοι. Αυτές οι κατανάθεσεις είναι κατοξιδότηση πράξης. Και η διαδικασία προβλέπει ότι εάν σε αναθεώρηση βρεθεί ασυμβατότητες θα πρέπει το κράτος μέλος να επαναδιαπραγματευτεί. Αν δεν τα καταφέρει το, κράτος, το συγκεκριμένο κράτος θα πρέπει να μπει στο πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποσυρθεί. Δίκτυα ασφαλείας τότε μόνο μπορεί να επικαλεστεί κανείς. Ο όποιος επομένως φοβάται για τις επενδύσεις θα πρέπει να σκεφτεί ότι πουθενά δεν υπάρχει απουσία κινδύνου, απουσία ρίσκου σε μια επένδυση. Άρα ελπίζουμε θα γίνουν βήματα πρόοδου, πάντως δεν έχουμε βρει την οριστική διατύπωση. Κύριε Στούτερ, σας ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρθηκε πολλέ φορέ στην ε, συζήτηση ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε τώρα πρέπει να δώσουμε το λόγο, εάν υπάρχει ο προσωπό για να μα πει τι γίνεται. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ του βουλευτέ για τι απόψει του που ήταν πάρα πολύ χρήσιμε και ενδιαφέρουσε. Πρόκειψε από τα όσα ακούσαμε ότι πρόκειψε ότι συμφωνείτε όσον αφορά τους στόχους του κανονισμού. Δηλαδή θέλω υπάρχει ε, επιδίωξη ασφαλής δικαίου και σταθερότητας για τους επενδυτές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειάζεται τα κράτη-μέλη να αγκαλιάσουν και να, φροντίσουν τα όσα θέλουμε να θεσπίσουμε. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονισμό που να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει σε περίπτωση προβλήματο. Και δίκιο κύριο Κάσπαρη. Ήδη έχουμε κάποια μέσα προβλέπει η συνθήκη. Δηλαδή την διαδικασία που παραβάσει όμω. Επίση έχει ο κύριο Σιλταρδίκιο εκεί που είπε ότι ίσω δεν είναι το και τόσο πρακτικέ αυτέ οι λύσει γιατί δεν προσφέρουν ασφαλεία δικαίου γιατί η, ασφάλεια, η προσφυγή επί δεν αφήνει περιθώρια σε περίπτωση προβλημάτων. Γι' αυτό και εμείς προτείναμε τα άρθρα 5 και 6 και είπαμε ότι έτσι θα μπορούμε να λάβουμε υπόψη και αυτές τις εκδοχές ε, στις ε, διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη ή τόσο με οποιονδήποτε και είπαμε ότι αυτόματα θα έρεται η έγκριση μετά από πέντε χρόνια. Αυτά να μην συνδεθούν μεταξύ τους, γιατί η αναθεώρηση υποτίθεται θα οδηγούσε σε έκθεση της Επιτροπής. Εκεί θα αποτυπωνόντουσαν τα προβλήματά μας. Τα οποία κατόπιν θα βλέπαμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα λύσουμε στο μέλλον. κάποια από αυτά τα μέτρα είναι το, τελευταίο καταφύγιο και ίσως ε, είναι αλήθεια ότι αυτό, η διατύπωση σε, αυτά τα δύο άρθρα που συζητούμε δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και ίσως χρειάζεται κάποιο χτένισμα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και ασφαλή δικαίωμα. Πέραν αυτών θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εμπλακεί σε περαιτέρω συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο. Και έτσι να δούμε τι συμβασμός μπορεί να εξευρεθεί. Και έτσι να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τους επενδυτέ, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την, τις πολιτικές μας. Ο πρόεδρος νομίζω ότι σε σημαντικά ε, σημεία Υπάρχει έδαφος για συμβασμό. Και ίσως θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα παραπέρα. Το χρονοδιάγραμμα τι προβλέπει. Ψήφιση της έκθεσης με 5-16 Μαρτίου θα προσπαθήσετε να βρείτε καινούργιε λύσεις οπότε μπορεί κάτι να αλλάξει. Ε, κύριε Πρόεδρε, μια που ήρθατε, μπορείτε να συνεχίσετε να προεδρεύετε Και εγώ σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πάβελ που με αντικαταστήσατε με τόσο κομψό τρόπο. Τώρα προχωρώ στο 13 αλλά πρώτα έχω να σας πω το εξής. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως των συντονιστών Τη 13 η Φεβρουαρίου έχουν διανεμηθεί και θα θεωρηθούν εγκεκριμένα στο τέλο τη συνεδρία εφόσον δεν προβληθούν ενστάσεις. Ε, αυτή η ανακοίνωση ήταν αναγκαίο να γίνει. Τώρα, ας προχωρήσουμε στο υπαριθμό 13 θέμα της ημερήσια διάταξης. εξέταση ερώτηση με έτοιμα προφορικής απάντησης σχετικά με τις ελεύθερε συναλλαγές με την Ινδία όπως έχουν αποφασίσει οι συντονιστές μας στι 7 Φεβρουαρίου που έχουν συντάξει ένα κείμενο ερώτησης σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ινδία. Το κείμενο σας έχει διανεμηθεί. αναμένεται η απάντηση ορισμένων πολιτικών ομάδων θα πρέπει να αποφασίσουμε πρώτα εάν θα ψηφίσουμε το κείμενο όπως έχει υποβληθεί ή αν θα δώσουμε προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών που θα ήταν η Τετάρτη Μαρτίου. ώστε η ψηφοφορία του κειμένου να γίνει στις 15 Μαρτίου. Φιέλνερ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε συμφωνήσει πλήρως. Γι' αυτό εκκρεμεί το θέμα. Ίσως υπάρχει περιθώριο συμφωνίας αλλά όχι στην βάση του υφισταμένου κειμένου. Ιδίω η παράγραφος 2 θα έπρεπε να τροποποιηθεί και εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος θα ζητήσω να τροποποιηθεί η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 ώστε να περιληφθεί και η βαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη που βασίζεται σε έρευνα διότι αναφέρουμε την ε, φαρμακευτική βιομηχανία φαρμάκων άνευ επωνυμία επωνυμίας και άλλα θέματα, αλλά δεν, δεν αναφέρουμε την φαρμακευτική βιομηχανία βασισμένη, την παραγωγή δηλαδή βασισμένη στην έρευνα. Έτσι θα τα περιλάβουμε όλα. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει όντω να δοθεί η δυνατότητα υποβολή τροπολογιών. Κύριε Σόλτ, άρα δεν θα ψηφίσουμε σήμερα. από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος άκουσα παρατήρηση να την απάνω υπόψη μου λέει ο κ. Σόλτς αλλά θα ήθελα να έρθω πάλι ε, στο σημείο 1 υπάρχει εκεί το λεγόμενο sustainable chapter είναι σημαντικό αυτό να μην έρθει μετά τη συνολική διαπραγμάτευση του κειμένου και να ψάχνουμε να βρούμε πού μπορούμε να βάλουμε τρεις-τέσσερις γραμμές για τα οικολογικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την βιωσιμότητα είναι σημαντικό είναι ένα θέμα σημαντικό τομής το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και στις διαπραγματεύσεις του κειμένου της ε, συμφωνίας. Θα μπορούσα να δεχθώ αυτή τη διατύπωση, αν όμως τελικώς αποφασίσουμε να υποβάλουμε πρόταση ψηφίσματος, θα πρέπει σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος να δώσουμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Πάντως κατά τα άλλα μπορώ να δεχθώ αυτό το συμβασμό για την ώρα. Άρα δεν υπάρχει, λέει ο Πρόεδρος, συμφωνία επί του κειμένου ως έχει. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι θα <clears throat> ανοίξουμε προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών μέχρι τις 4 Μαρτίου στις 6 το βράδυ, το απόγευμα. και μετά δεν έχουμε άλλα. Θα προχωρήσουμε τώρα στην ε, συνεδρία των συντονιστών. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν είναι συντονιστές ή πρόσωπα που επιτρέπεται να παραμείνουν στη συνεδρία των συντονιστών, παρακαλώ λοιπόν τα πρόσωπα αυτά να εξέλθουν τις αιθούσεις ησύχως. Μόνο συντονιστές γραμματεία, νομική υπηρεσία, οι αξιωματούχοι των πολιτικών ομάδων και οι συνεργάτες των συντονιστών. Μόνο αυτοί επιτρέπεται να παραμείνουν.